Bene. Cari colleghi, dobbiamo credo cominciare perché il signor Ξεκινάμε. Ο Υπουργό είναι μαζί μα και έχουμε μια ημερήσια διάταξη αρκετά βεβαρημένη. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Υπουργό Μαρτώνη, Υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας, προεδρεύοντα του Συμβουλίου, ο οποίος δέχτηκε την πρότασή μας και θα μας μιλήσει και για τη διαδικασία διεύρυνσης στο πολιτικό πλαίσιο των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ουγγρική Προεδρία, ιδιαίτερα εσάς κύριε Υπουργέ, για το δυναμισμό και την ενέργεια που δώσατε στην διαδικασία της διεύρυνσης και για την Κροατία ιδιαίτερα έχει φτάσει σε μια φάση πλέον πάρα πολύ κοντινή στην κατάληξη των διαπραγματεύσεων είδαμε ποια ήταν και η ανακοίνωση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υπάρχουν όλα τα κεφάλαια πλέον ανοιχτά και είναι στην τελική φάση. Μια άλλη υποψήφια χώρα είναι η Ισλανδία. Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να αποφασιστεί να ξεκινήσουν και με αφορμή την διακυβερνητική της 27 Ιουνίου. σκεπτόμαστε να κλείσουμε δύο από τα κεφάλαια και να ανοίξουμε τα υπόλοιπα. Ίσως ένα θέμα το οποίο έχει βρεθεί λίγο στη σκιά τον τελευταίο καιρό είναι η Τουρκία γιατί επανερχόμεθα συχνά στα ίδια πράγματα και καλό θα είναι υπό το φως και των τελευταίων εκλογών βέβαια στην Τουρκία να σας ακούσουμε κύριε Υπουργέ για τις εκτιμήσεις που κάνετε. Δεν θέλω να χάσουμε άλλο χρόνο. Το θέμα είναι να μην ακούει κανείς αυτά που λέω εγώ, αλλά τις δικές σας σκέψεις και χωρίς περαιτέρω πολυσιεργία σας δίνω το λόγο και θα σας ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση, τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για χαρά σε έναν βαθμό. Τώρα να είμαι σε θέση να σας παρουσιάσω σήμερα τις εξελίξεις των τελευταίων 5,5 μηνών στον τομέα της διεύρυνσης και να αναπτύξω κάποια σχετικά θέματα στον τομέα. Πριν από πέντε μήνες ήμουν πάλι εδώ και αν θυμάμαι καλά είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρει η διεύρυνση εν γέννη και σε σχέση με τις επιμέρους χώρες. Σας είχα επίση μιλήσει για το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας και τις προτεραιότητές μας. Ιδιαίτερα δεν είχα υπογραμμίσει το γεγονός ότι μια από τις προτεραιότητες του προγραμματός μας είναι η πρόθεση της διαδικασίας διεύρυνσης. Πιστεύω δεν αμφισβητεί κανείς το γεγονός ότι η διεύρυνση έχει στρατηγική σημασία. Ενισχύει την Ευρώπη σε όρους οικονομικούς όσο και πολιτικούς. Θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπον αξιόπιστο. Και ταυτόχρονα πρέπει να διεξάγεται με βάση όλα τα κριτήρια της διεύθυνσης που έχουν προβλεφθεί και που θα πρέπει να πληρούνται κατά τον ίδιο τρόπο από όλες τις υποψήφιες χώρες. Το σύνθημα της Ουκρικής Προεδρίας ήταν η ε, ε, ισχυρή Ευρώπη. Και στο σύνθημα αυτό εγγράφηκε και οι προσπαθίες μας για τη διεύθυνση. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να υπογραμμίσω ότι μια Ευρώπη διευρυμένη, μια Ευρώπη ανοιχτή, είναι ασφαλώς ισχυρότερη με καθένεια από μια Ευρώπη που θα έχει τις πόρτες σφαλισμένες στον εξωκόσμο και που θα ασχολείται μόνο με τα εσωτερικά της προβλήματα. Ταυτόχρονα είπαμε εξ αρχής, αλλά τώρα το πιστεύω ακόμη περισσότερο, ότι είναι μια διαδικασία η διεύρυνση. Πρέπει να παρουσιάζει συνέχεια. Και άρα κάθε μία προεδρία θα πρέπει να στηρίζεται και να αναπτύσσει το έργο, να στηρίζεται στο και να αναπτύσσει το έργο της προηγούμενης. συνεχίζουμε το έργο των προηγούμενων προεδριών και παραδίδουμε στο προσεχές τρίο Πολωνία, Δανία, Κύπρο που θα συνεχίσει το έργο μας. Αυτό το λέω γιατί δεν πιστεύω σε έπαθλα, δεν πιστεύω σε τρόπαια, δεν πιστεύω στο να διεκδικεί κανείς δάφνες για το τι έπραξε, τι δεν έπναξε, τι επέτυχε κτλ. Πιστεύω όμως ότι πρόκειται για μια διαδικασία, μια διαδικασία που αποβαίνει στο συμφέρον όλων μας, πάνω απ' όλα συμφέρον της Ευρώπης μια διαδικασία στην οποία κάθε μια Προεδρία έχει πολύ απλή, ένα πολύ απλό μερίδιο της δουλειάς, να κάνει τη δουλειά της δηλαδή και να προωθήσει τη διαδικασία. Τρίτο στοιχείο. Συμφωνώ με όλοι, το είπα και νωρίτερα. με μια διαδικασία αξιόπιστη η οποία σημαίνει και διατύπωση απαιτήσεων και παροχή αποτελέσματος, παραγωγή αποτελέσματος. Αυτά δύο Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εφόσον τα ορόσημα τα επιτυγχάνει κανείς, τα φτάνει κανείς, τότε Φυσικά κατά κύριο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταγράψει τις εξελίξεις και τα γεγονότα αλλά και εμείς από πλευράς μας πρέπει να δώσουμε τη σωστή απάντηση, την αναμενόμενη απάντηση. Και θα ήθελα προκαταρκτικά επίσης να επισημάνω ότι η κέρια σημασίας παράγων είναι η καλή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Από την εμπειρία μας αυτό το εξάμεινο βλέπουμε ότι στον τομέα της διεύρυνσης η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων έχει προχωρήσει κατά τρόπο εξαίρετο και χωρίς καμιά επιφύλαξη πάνω να το πω αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε καταπληκτική δουλειά, καταπληκτική ε, μεγάλη πρόοδο, ιδιαίτερα στους τελευταίους μήνες και όσον αφορά το θέμα της Κροατίας, το οποίο θα επανέλθω σε λίγο. Επίσης, η πολιτική υποστήριξη που προσφέρθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν και είναι πάρα πολύ σημαντική. Το Συμβούλιο συνεργάστηκε με την, με την Επιτροπή. Η Προεδρία φυσικά αποδίδει τεράστια σημασία στην ε, αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας. Και αν υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στο θέμα αυτής της διεύρυνσης σε μεγάλο βαθμό πιστεύω οφείλονται και θα πρέπει να αποδοθούν σε αυτή την απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Με αυτές τις προκαταρκτικές λοιπόν παρατηρήσεις επιτρέψαμε τώρα να περάσω εν συντομία στα γεγονότα. Και να εκθέσω τα επιτεύγματά μας. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει, όταν λέω εμεί, ε, μα δεν εννοώ την Ειδική Προεδρία, εννοώ όλων μα τα επιτεύγματα. Και ξεκινώ με το ερώτημα. Έχουμε προχωρήσει στο θέμα της διεύρυνσης τώρα περισσότερο από ότι ε, έχουμε σε ένα σημείο πιο προχωρημένο από ό,τι ήμασταν πριν από έξι μήνες. Έχουν ε, ε, πραγματοποιηθεί ουσιαστικά βήματα πρόοδου. Είναι σε καλύτερη κατάσταση τώρα η διαδικασία της διεύρυνσης από ό,τι ήταν πριν από έξι μήνες. Θα πρέπει για να δώσουμε απάντηση να περάσουμε στην εξέταση των επιμέρους υποψηφίων χωρών. Αλλά πριν ξεκινήσω θα πρέπει να παρατηρήσω ότι η διεύρυνση είναι ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, είναι μια σύνθετη δραστηριότητα και ασφαλώς οτιδήποτε συμβαίνει στην, ε, υποψηφ... στην ε, περίπτωση μιας υποψήφιας χώρας έχει άμεσες επιπτώσεις και στην περίπτωση μιας άλλης υποψήφιας χώρας. Άρα ε, δεν μπορούμε να τα δούμε αυτά αποκομμένα. Και μιλούμε γενικά για την διαδικασία της διεύρυνσης, αλλά και για τα δυτικά, ε, περισσότερο για τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και για υποψηφίες χώρες όπως η Τουρκία. Στο θέμα των Δυτικών ε, Βαλκανίων όμως ξέρουμε ξεκάθαρα ότι η επιτυχία ή η αποτυχία μιας συγκεκριμένη χώρας στην πορεία της για την ένταξη έχει άμεση επιπτώσεις στην διαδικασία προσχώρησης όλων των κρατών. Ε, εάν επιτύχει μπορεί να δώσει μια νέα πνοή στη διαδικασία, εάν αποτύχει μπορεί να συμπαρασύρει, γιατί υπάρχει αυτή η ψυχολογική στάση απέναντι στην ε, πιθανότητα της διεύρυνσης, η οποία δεν υπάρχει μόνο στην ευρωπαϊκή πλευρά, υπάρχουν συναισθήματα τέτοιας φύσεως και ε, σε επίπεδο κρατών, υποψηφίων κρατών, που σημαίνουν ότι ανάλογα με την επιτυχία ή την αποτυχία μιας διαδικασία μπορεί να επηρεαστεί συνολικά η ψυχολογική διάθεση και η στάση απέναντι στη διεύρυνση στις χώρες αυτές. Η Κροατία μας έχει απασχολήσει καταρχάς τους τελευταίους έξι μήνες ιδιαίτερα. Πρόοδο σημειώνουμε. Ήδη προσημειώσαν οι προηγούμενες προεδρίες όπως σας γνωρίζετε. Η Βελγική Προεδρία ολοκλήρωσε δύο κεφάλαια στους τελευταίους μήνες. Μετά εμείς ολοκληρώσαμε, κλείσαμε τρία κεφάλαια. Γεωργία, περιφερειακή πολιτική και πιο πρόσφατα την αλία Μας μένουν τέσσερα κεφάλαια και δύο εβδομάδες χρόνος. Αλλά έχουμε φτάσει σχεδόν πλέον στην ε, γραμμή του τερματισμού και χωρίς να θέλω να προδικάσω τις εξελίξεις, έχουμε μπει πλέον στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων. Ξέρετε πολύ καλά τι συνέβη στις 10 Ιουνίου, θα διαβάσατε όλοι φαντάζομαι τις δηλώσεις του Προέδρου Μπαρόσο, του κυρίου Φίλε. Η κατάσταση επομένω σας είναι γνωστή. Συνεχίζονται οι συζητήσεις εντατικά Και θα ήθελα να υπογράψω για μια άλλη μια φορά το τεράστιο έργο που έχει επιτελέσει η Ευρωπαϊκή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε τα τελευταία τέσσερα σχέδια κοινών θέσεων. Πολύ καλή δουλειά. Και μάλιστα με πολύ ταχύς ρυθμούς. Γνωρίζετε τα συμπεράσματα αυτών των σχεδίων θεωρείται ότι ε, πλέον πληρούνται οι προϋποθέσεις ή επαρκώς πληρούνται οι προϋποθέσεις. Επαρκώς σημαίνει ότι αρκεί. Άρα είναι σε το συμπέρασμα, εν προκειμένου. Μας μένει να διευκρινίσουμε ορισμένα ζητήματα που μας απασχολούν τα επεξεργαζόμαστε με εντατικούς ρυθμούς. Είμαστε αισιόδοξοι όπως ολόκληρο το εξάμεινο. Ε, Διατηρήξαμε την ε, αισιοδοξία μας έστω και σε περιόδους όπου δεν υπήρχαν πολλοί λόγοι για αισιοδοξία. Εμεί δεν ε, αλλάξαμε στάση, παραμένουμε αισιόδοξοι λοιπόν και έτσι μπορώ να σας πω σήμερα ότι ελπίζουμε και υπάρχουν σαφείς προσδοκίες πώς θα μπορέσουμε να κλείσουμε όλα τα κεφάλαια και την διαδικασία των διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός. Σημαντικές συνεδριάσεις προβλέπονται για τις 21 Ιουνίου με το Συμβούλιο των Κοινωνικών Υποθέσεων το οποίο θα μπορούσε να συστήσει τα ακόμη εκκρεμή ζητήματα συζήτηση επί της ουσίας δηλαδή και Στη συνέχεια οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μπορούν στις 23 και 24 να ασχοληθούν με το ζήτημα και έχουμε και τη δυνατότητα για μια διακυβερνητική μετά από αυτό μέχρι τα τέλη Ιουνίου τελευταία ημέρα της Προεδρίας, 30 Ιουνίου, όπως γνωρίζετε, δεν μπορεί να γίνει ε, διάσκεψη για προσχώρηση στις 31 Ιουνίου, γιατί δεν υπάρχει 31 Ιουνίου. 30 Ιουνίου είναι η τελευταία μας μέρα λοιπόν και στις 12 το μεσάρχη της 30 Ιουνίου πρέπει να έχουμε κλείσει την υπόθεση. Είναι δυνατόν καλύτερα να έχουμε κλείσει την υπόθεση. Θα ήθελα να υπογράψω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για μια διαδικασία. Δεν έχει να κάνει με... Ε, έπαθλα, με τρόπεα, με δάφνες. Έχει να κάνει με το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βεβαίως και τα συμφέροντα του υποψηφίου κράτους. Και όπως είπα και νωρίτερα, οτιδήποτε και να συμβεί στη διαδικασία της διεύρυνσης και ανεξάρτητα της, ε, του ποια είναι η υποψήφια χώρα, έχει αυτό επιπτώσεις στην, στο σύνολο των υποψηφίων κρατών. Αυτό νομίζω το βλέπουμε ήδη ξεκάθαρα. Στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κροατία να αντανακλάτε, βλέπουμε δηλαδή ότι χάρη στην επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας ένταξης της, προ... της Κροατίας υπήρξαν και άλλες χώρες και άλλες διαδικασίες που επίσης αναζωογονούνται λέω πράγματα βέβαια γνωστά σε όλους αλλά είναι σοφές ότι όλες οι υποψηφιέ χώρες με μεγάλη προσοχή παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στην Κροατία. Αν δεν κοιτάξουμε την περίπτωση της Σερβίας, είναι σαφές ότι και εκείνοι έχουν δώσει μεγάλη όθηση στη δική τους διαδικασία προσχώρησης, όπως άλλωστε και άλλες χώρες, που δίνουν δείγματα επιτάχυνσης, δείγματα λήψης των πολιτικών αποφάσεων που χρειάζονται για να προχωρήσει η διαδικασία. είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε η μαγεία της διαδικασίας της προσχώρησης, δηλαδή η ενέργεια, η δράση αυτή της εξέλιξης στην ε, υποψηφιότητα μίας χώρας μεταδίδεται στις υπόλοιπες χώρες που παίρνουν το σωστό μήνυμα και αντιδρούν αμέσως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό Και γι' αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όταν μιλούμε για μια συγκεκριμένη χώρα, μιλούμε για μια περιοχή περισσότερο παρά για ένα κράτος μόνο. Θα ήθελα λοιπόν και άλλη μια φορά να υπογραμμίσω πως όλοι έχουμε ενδιαφέρον να προωθήσουμε την διαδικασία της προσχώρησης. Πρέπει βέβαια να πιστεύουμε σε αυτή τη διαδικασία προσχώρησης. υπάρχει και δεν πρέπει να το ε, γνωρίζουμε αυτό και το φαινόμενο της κόπωσης ε, σε σχέση με τη διεύρυνση της υπερβολικής δηλαδή ανασχόλησης και τελικά αρνητικής αντίδρασης στη διαδικασία της διεύρυνσης. Αυτό μπορεί να, μας, ε, να εμφανιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο επίπεδο των υποψηφίων κρατών. Υπάρχει δηλαδή ψυχολογικός παράγον, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να υπογραμμίσω ότι η διεύρυνση έχει μεγάλη σημασία για όλους μας, διότι ε, ζούμε σε εποχές γεμάτες προκλήσεις και εάν δεν έχουμε αυτοπεποίθηση δεν μπορούμε και να εμφανιστούμε αξιόπιστοι έναντι των λοιπόν, έναντι του έξω κόσμου. Κύρια δε, προϋπόθεση για την επιτυχία μιας ε, διαδικασίας διεύρυνσης είναι η αυτοπεποίθηση από πλευράς μας και η εμπιστοσύνη σε αυτή τη διαδικασία διεύρυνσης. Για να προχωρήσω τώρα στο θέμα των εξελίξεων το τελευταίο εξάμεινο, που είναι σαφής νομίζω στην περίπτωση της Κροατίας. Η πρόοδος είναι δεδομένη, δεν αμφισβητείται. Ό,τι και να συμβεί σε επόμενες δύο εβδομάδες ε, δεν αμφισβητείται η πρόοδος που σας περιέγραψα εν συντομία. αλλά θα μπορούσα να προχωρήσω για να παρουσιάσω τα θέματα αναχώρα και αν εξετάσουμε όλες τις χώρες, τουλάχιστον στις περισσότερες υποψήφιες, ή που χώρες που έχουν υπο... βάλει αίτηση για υποψηφιότητα, ε, υπάρχει πρόοδος. Μίλησα λοιπόν για την Κροατία, αλλά πέραν αυτής έχουν και οι άλλες χώρες σημειώσει τη δική τους πρόοδο η καθεμία. Ανέφεραν όλοι τη Σερβία, Φερπίν. Και εκεί υπάρχει κινητικότητα. Και αυτή δεν την αποδίδω μόνο στη σύλληψη και την ε, ε, μεταφορά στη Χάγη του στρατηγού Μλάντιτς. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Υπάρχει ένα κλίμα πιο φιλοευρωπαϊκό στη Σερβία. Εν γέννη. Το βλέπουμε και στην ε, πολιτική ελίτ αλλά και σε μεγάλα τμήματα του λαού. που αισθάνονται δυσφορία για το παρελθόν και λόγω των εξελίξεων και το διάλογο μεταξύ Πρίστινα και Βελιγραδίου. που καλύπτουν θέματα σε τεχνικό ακόμη επίπεδο, γιατί χρειάζεται ακόμη να ληφθούν και οι πολιτικέ αποφάσει, αλλά γίνονται σε τεχνικό επίπεδο και υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, πρόοδο σε θέματα όπω οι τηλεπικοινωνίε, όπω το κτηματολόγιο, όπω η εγγραφή στα Μητρώα των Πολιτών, η ελευθερία διακίνηση. Εκεί έχει σημειωθεί πρακτική πρόοδος και πιστεύω ότι τουλάχιστον από την ε, δική μας πλευρά μπορούμε να αποδώσουμε σε μεγάλο βαθμό τις προόδους αυτές στις ε, ευρωπαϊκές προοπτικές που έχουν ανοίξει και που διευκολύνουν τις συζητήσεις αυτές. Μαυροβούνιο. Άλλο ένα προφανές παράδειγμα. Έχει δοθεί το καθεστώς του ψηφίου κράτους στο Μαυροβούνιο ακόμη πολλή δουλειά έχουν μπροστά τους. σε 7 κυρίως τομείς. Τώρα ετοιμάζουν ένα σχέδιο προγράμματος δράσης υπό την καθοδήγηση του ε, Πρωθυπουργού τους. Και... Με αποτέλεσμα και σαν αποτέλεσμα μάλλον της εφαρμογής αυτού του προγράμματος δράσης και επί τη βάση της αξιολογήσεως βέβαια την οποία θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και μπορεί να δοθεί ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών γιατί φυρών ΦΥΡΟΜ είναι υποψήφια έξι χρόνια περίπου οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν μπορέσει να ξεκινήσουν ακόμα όπως ξέρετε υπάρχει μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές σε δύο πλευρές για το θέμα του ονόματος. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε την άποψή της, η οποία όμως δεν ακολουθήθηκε από τα κράτη-μέλη. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί ομόφωνα από τα κράτη-μέλη για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Όπως γνωρίζουμε τώρα πλέον, οι συζητήσεις συνεχίζονται και από ό,τι ακούμε και από τις δύο πλευρές έχει υπάρξει μια γυτνίαση των θέσεων των δύο πλευρών, δεν ξέρω πόσο κοντά είναι, αλλά πιστεύουμε ότι Η σύγχρονη γεωμετρία δείχνει ότι ακόμα και οι παράλληλες γραμμές σε κάποια φάση μπορεί να συναντηθούν. Οπότε ελπίζουμε ότι ακόμα και αν υπάρχουν διαφορές κάποια στιγμή θα εξομαλυνθούν. Τώρα μιλώ για τη χώρα μου. Εμείς έχουμε κάθε συμφέρον οι διαπραγματεύσεις αυτές να ρυθμιστούν και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μετά από την πρόταση και του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέγουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη ΦΥΡΟΜ. Αν φύγουμε από την περιοχή αυτή για λίγο, αν και εγώ πρέπει να περιοριστώ στις υποψήφιες ή σχεδόν υποψήφιες χώρες, έχουμε τη διαδικασία διεύρυνσης με την Τουρκία. Αυτό είναι ένα μέγιστο στρατηγικό πρόβλημα. Είναι σαφές ότι δεν ξεκίνησε κάποιο νέο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας και δεν ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο ούτε και κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας και δεν έχω πολλές ελπίδες ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο εβδομάδες. Γιατί το να ξεκινήσουν, εν πάση περιπτώσει, οι συζητήσεις σε κεφάλαια, αυτό εξαρτάται από τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ είχα μιλήσει για την Τουρκία και παλαιότερα και είχα πει ότι σύμφωνα με τη θέση μας έχει κάθε στρατηγικό συμφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία και είχα πει επίσης ότι σε πρακτικό επίπεδο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα επιπλέον βήμα αναγνωρίζοντας πάντα τις δυσκολίες που έχει η διαδικασία. Αλλά είχαμε εκφράσει την ελπίδα ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση του 8ου κεφαλαίου για τον ανταγωνισμό. Ήταν η ελπίδα μας. Δεν τα καταφέραμε. Για την Τουρκία η περίοδος που πέρασε ήταν πολύ ιδιαίτερη θα έλεγα, ήταν προεκλογική περίοδος, έγιναν οι εκλογές την προηγούμενη εβδομάδα. Στις 12 Ιουνίου Αυτό λέω και εγώ. Ο κ. είπε την προηγούμενη Κυριακή. Ναι, ναι, συμφωνούμε, υπάρχει ομοφωνία για την ημερομηνία τέλεσης των εκλογών. Όλοι πιστεύουμε και θα ήθελα να αναφερθώ και στις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο πρόεδρος Μπαρόσο και ο πρόεδρος Βαν Ρομπάι. Και οι δύο εξέφρασαν την ελπίδα οι εκλογές αυτές να δώσουν μια νέα όθηση στην διαδικασία όχι μόνο γενικότερα στη διαδικασία εξυγχρονισμού των θεσμών γενικότερα στη χώρα αυτή, αλλά να δώσουν και μια νέα όθηση στις διαπραγματεύσεις ε, για την ένταξη της Τουρκίας. Τα δύο αυτά θέματα φυσικά συνδέονται. Θα ήταν δύσκολο να περιμένει κανείς από την τουρκική κυβέρνηση να κάνει τεράστιες αλλαγές στον τομέα των επιδοτήσεων, στον τομέα του ανταγωνισμού, της πολιτικής ανταγωνισμού, των ομοθετικών ρυθμίσεων για τον ανταγωνισμό πριν τις εκλογές. Τώρα όμως άλλαξε η κατάσταση και ελπίζουμε ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν μόνο τρία καταρχάς κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να ανοίξουν. Δεν θέλω να υποτιμήσω α, τις πολιτικές δυσκολίες που οδηγούν στο να έχουν μπλοκαριστεί πέντε συν έξι κεφάλαια, 11 συνολικά. Ταυτόχρονα όμως όλοι γνωρίζουμε ότι αυτές οι πολιτικές δυσκολίες και τα προβλήματα θα πρέπει να επιληθούν γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει ουσιαστική προόδος στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Να φύγω τώρα από την Τουρκία, Ισλανδία. Έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Θα τεθεί το θέμα στη διακυβερνητική της 27ης Ιουνίου Θα ανοίξουμε τέσσερα κεφάλαια. Και ελπίζουμε δύο από τα τέσσερα αυτά κεφάλαια να κλείσουν άμεσα στα πλαίσια αυτής της συνάντησης. Το 25 για την έρευνα και το 26 για τον πολιτισμό και την παιδεία. Βέβαια αυτά είναι τα λεγόμενα εύκολα κεφάλαια. Νομίζω το ίδιο κάνουμε και σε άλλες περιπτώσεις με άλλες χώρες όταν διαπραγματευόμεθα. Αλλά θα υπάρξουν κάποια πιο ακανθώδη προβλήματα όσο προχωράμε. Τα ξέρετε τα προβλήματα αυτά. Δεν θέλω να τα απαριθμίσω, δεν θέλω να περάσω τώρα σε λεπτομέρειες. Να αναφερθώ σε μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη η αρχή εποπτείας της ΕΖΕΣ η οποία εξέδωσε μία ανακοίνωση χτες ή προχθές για την υπόθεση iSave. Ελπίζουμε το θέμα αυτό να προχωρήσει σε μια κάποια λύση όσο προχωράνε και οι διαπραγματεύσεις. Εδώ υπάρχουν λοιπόν κάποιες εκκρεμότητες. Πάντως μπορούμε να είμαστε, έχω την αίσθηση αισιόδοξη για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων αυτών με την Ισλανδία. Τώρα στις χώρες που θα ήθελα να είναι υποψήφιες, που δεν είναι ακόμα υποψήφιες, αναφέρθηκα ήδη σύντομα στη Σερβία. Πολλά θα εξαρτηθούν από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής το μήνα Οκτώβριο. Οι Σέρβοι είναι τώρα αρκετά αισιόδοξοι και περιμένουν όχι μόνο να τους δοθεί το καθεστώς της υποψήφιας χώρας, ελπίζουν να υπάρξει και ημερομηνία για την κίνηση των διαπραγματεύσεων. Αυτό τώρα είναι μια εκκρεμότητα βέβαια, δεν θέλω να το σχολιάσω θα ήθελα να πω ότι από ουγγρικής πλευράς υποστηρίζουμε πλήρως την Σερβία στις δικές της φιλοδοξίες έχουμε εθνικά συμφέροντα θα έλεγα είναι γειτονική χώρα περιφερειακά συμφέροντα και ελπίζω ότι ακριβώς γι' αυτό όταν ολοκληρωθούν σύντομα ελπίζω οι διαπραγματεύσεις με την Κροατία η επόμενη στη σειρά είναι η Σερβία κατά τη γνώμη μας και πρέπει να βοηθήσουμε τη διαδικασία αυτή με τη Σερβία όσο μπορούμε. Έχουμε βέβαια τρεις άλλες δύσκολες περιπτώσεις. Δεν θα μπω από εδώ και πέρα σε λεπτομέρειες γιατί δεν ανήκουν θα έλεγα τα της διεύρυνσης προς το παρόν αφορούν γενικά την, τα Βαλκάνια, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Αλβανία και ε, Σχετικά με το κοσυφοπέδιο έχουμε να κάνουμε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Αναφέρθηκα στον διάλογο ο οποίος συνεχίζεται ανάμεσα στην κυβέρνηση της Πρίστινα και στην κυβέρνηση του Βελιγραδίου. Είναι πολλά υποσχόμενος ο διάλογος αυτός. Για τις άλλες δύο χώρες υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν προκλήσεις. Δεν θα τις τώρα. Τώρα αν μου θέσετε ερωτήσεις προφανώς θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ. Μπας περιπτώσει τώρα για να κλείσω λίγο. Πρώτον, έχει υπάρξει πρόοδος με τις περισσότερες υποψήφιες και φιλοδοξούσες να γίνουν υποψήφιες χώρες. Η Κροατία είναι μπροστά και εφόσον πράγματι επιβεβαιωθεί η επιτυχία της διαδικασίας στο τέλος Ιουνίου θα επηρεάσει νομίζω θετικά το σύνολο της περιοχής και τις διαδικασίες ένταξης των υπολείπων. Και δεύτερο σημείο είναι ότι σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια η κατάσταση είναι άνηση θα έλεγα και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των υποψηφίων χωρών. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία αστάθειας, κινδύνων Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Μέχρι τώρα υπογράμμιζα τις θετικές πλευρές, θα έλεγα, αυτών των διαδικασιών, κυρίως της Κροατίας. Υπάρχουν όμως και αρνητικές πλευρές. Είναι ο κίνδυνος, οι απειλές οι οποίες υπάρχουν σε κάποιες χώρες της περιοχής. Δεν θα πρέπει να πιστεύουμε ότι όλες οι δυσκολίες που είχαν αυτές οι χώρες έχουν τώρα ξεπεραστεί και ότι το μέλλον είναι εξασφαλισμένο για όλες αυτές τις χώρες. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στα πλαίσια της διαδικασίας διεύρυνσης. Τελευταία λέξη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν και πόσο πολύ βοήθησαν τους τελευταίους 5,5 μήνες Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είχε ένα ρόλο κλειδί στην περίπτωση της Κροατίας αλλά και γενικότερα. Σας είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που έκαναν πάρα πολλά και το αναγνωρίζω. Να αναγνωρίσω τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες αναντικατάστατος και φυσικά όλες τις χώρες οι οποίες συνεργάστηκαν υπήρξε πνεύμα συνένεσης, συνεργασίας ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες και τις τελευταίες μέρες είμαι σίγουρος ότι αυτό το πνεύμα συνεργασίας και συνένεσης θα συνεχίσει. Και στο τέλος της Προεδρίας μας θα μπορέσουμε να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με την Κροατία και ότι η διαδικασία διεύρυνσης θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί αξιόπιστα, με ασφάλεια και χωρίς κινδύνους. Ευχαριστώ Υπουργέ για μια πληρέστατη παρουσίαση. Θα δώσω το λόγο τώρα πρώτα στον κύριο Σβόμποντα, εισηγητής για την Κροατία, όχι πάνω από τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την εισαγωγή σας. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί δεν έχω πολλά να προσθέσω. Καταρχήν θα ήθελα να εκτιμήσω το έργο της Ουγγρικής Προεδρίας και την προσωπική σας δέσμευση στην περίπτωση της Κροατίας. Ίσως θα πρέπει να σταματήσετε το ρολόι στις 30 Ιουνίου έτσι όπως έγινε με την Αυστρία αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα ήταν ένα πετυχημένο τρόπο να ασχοληθούμε με αυτό. Βεβαίω τα αποτελέσματα είναι καλά, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την εφαρμογή και η διαδικασία παρακολούθησε μετά την είσοδο, μετά την προσχώρηση είναι σημαντική και μπορούμε να υποσχεθούμε στην Κροατία ότι αυτή τη στιγμή λάβουμε τα έγγραφα στο Κοινοβούλιο θα υπάρξει μια προσεκτική μεν, αλλά ταχεία διαδικασία για να ολοκληρωθεί. Προσεκτική βεβαίω, γιατί ξέρετε ότι μεταξύ του πληθυσμού σε ορισμένε χώρε υπάρχουν ορισμένε αντιδράσει, αντιστάσει και αμφιβολίε. Αλλά συνολικά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό και το Κοινοβούλιο αυτό θα συνεχίσει να υποστηρίζει τι φιλοδοξίε τη Κροατία. Δεύτερον, για τη Σερβία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπατε και θα ήθελα να τονίσω και να αναφέρω γιατί καμιά φορά το ξεχνάμε και με την Κροατία δώσαμε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας ακόμα και όταν όλα δεν είχαν επιληθεί. Βεβαίως δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις αλλά όπως βλέπουμε στην αρχή περίπτωση της Μακεδονίας πριν ε, υποβάλει υποψηφιότητα και πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αλλά ε, στην ε, Σερβία έχουμε τις εθνικιστικές δυνάμεις από τη μία και τις δημοκρατικές δυνάμεις από την άλλη, τις οποίες θα πρέπει να αποστείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, να συνεχίσουν την προσπάθειά τους και να έχουν μια θετική απάντηση από την Ευρώπη. Ε, εσείς θα παραμείνετε μεταξύ των, του Σώματος των Υπουργών Εξωτερικών και παρακαλώ να μείνετε στο ζήτημα της Σερβίας. Δεν μπορούμε βεβαίως να μειώσουμε το τις προποθέσει, αλλά θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι προ όλε τι χώρε και να αποστείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα ε, στην κρατία νέα, αλλά να μην ξεχνάμε και τι υπόλοιπε χώρε. αυτή θα ήταν μια εσφαλμένη τοποθέτηση και για να κερδίσουμε χρόνο θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ κύριε Σκουκάν, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις ανάμεσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και... και ποιο? Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Ε, ορίσατε και σας ευχαριστούμε για τα εισαγωγικά σας λόγια. Όταν η Ουγγαρία ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχαν κάποιες θεμητέ προσδοκίε θεμητές προσδοκίες ότι θα αναλάβει ενεργό ρόλο η Ουγγαρία στα Δυτικά Βαλκάνια δεδομένη της εμπειρίας και της εμπειρογνωμοσύνης αυτής της χώρας από την συνεργασία με τις χώρες αυτής της περιοχής. Και θα ήθελα να εκτιμήσω το έργο το οποίο επετέλεσε η Ουγγρική Προεδρία γιατί πραγματικά σηματοδοτεί ε, θετικά τις εξελίξεις στην περιοχή αυτή. Δύο στοιχεία θα ήθελα να τονίσω. Αυτό που είπατε κύριε Υπουργέ, ότι η επιτυχία ή η αποτυχία κάθε επιμέρους χώρα στην περιοχή που αφορά την διαδικασία της διεύρυνσης έχει θετικό ενδικό αντίκτυπο και στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Και αυτό έχει αποδειχθεί από την Κροατία, γιατί βεβαίως ο χρόνος έχει μία σημασία και θα ήταν ε, σωστό να... και θα πρέπει να υπάρξει, είναι σωστό να υπάρξει θετικός αντίκτυπος στις άλλες χώρες της περιοχής. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ και χαίρομαι που πραγματικά υλοποιείται είναι ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αποβούν αποτελεσματικά και να περάσουν θετικά τις μελλοντικέ εξελίξεις της περιοχής προς την Ευρώπη. Ε, εάν μιλούμε με μία φωνή όταν αποστέλουμε τα μηνύματα στις επιμένους χώρες ή στην περιοχή, θα πρέπει να μιλούμε ομόφωνα. Ε, αυτό δεν είναι εύκολο. Ορισμένε φορέ είναι δύσκολο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένη τη πολιτική του σύνθεση και των άλλων πολιτικών ε, τέρων στι ε, χώρε. Αλλά δεν υπάρχει άλλο τρόπο να πειράσουμε θετικά τι εξελίξει, γιατί εδώ βρίσκονται γιατί τα συμφέροντα μάλλον των χωρών και των πολιτών των χωρών αυτών θα πρέπει να αποτελούν την προτεραιότητα για όλους. Συμφωνώ μαζί σας ότι η διεύρυνση συνιστά μια πολύπλοκη, περίπλοκη διαδικασία, έχει διάφορα χαρακτηριστικά, διάφορες πτυχές και συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι υπάρχουν ορισμένες θετικές εξελίξεις αλλά και ορισμένα εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά εάν ε, δούμε τις προηγούμενες έξι τους προηγούμενους έξι μήνες ε, ε, πιστεύω ότι ένας ε, πιστεύω ότι το μέλλον της Κροατίας θα επηρεάσει θετικά την κατάσταση και η πρόοδος που σημείωσε το Μαυροβούνιο και η Σερβία ακόμα και στην περίπτωση της Βοσνίας Αρτσικοβίνης υπάρχει μια χτίδα φωτός, ελπίδας όταν δούμε τις πρόσφατες εξελίξεις. Ε, η Αλβανία είναι δύσκολη, όλοι το γνωρίζουμε, Υπάρχει, έχουμε τη διακοινοβουλευτική συνάντηση μαζί τους. Ε, δεν επιτάθηκαν πολλά, ειλικρινά, αλλά για πρώτη φορά έλαβε χώρα ένας ε, σωστός διάλογος χωρίς αμοιβέ προσβολές, επιθέσεις κλπ. Και σίγουρα αυτό θα είναι χρήσιμο. Ο κύριος Πρόεδρος μου ρίχνει ορισμένες ματιές, γι' αυτό θα σταματήσω. Ευχαριστώ. Λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε όλους να πάρουν το λόγο. Εσείς σαν πρόεδρος αντιπροσωπείας είχατε λίγα λεπτά περισσότερο, αλλά ας μην υπερβάλλουμε. Βάγγελ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μαρτώνη, είμαι πεπισμένος ότι η Ουγγαρία χρήζει σεβασμού για τα όσα έπραξε και για τα όσα πράξατε εσείς ο ίδιος προσωπικά για να κρατήσετε, διατηρήσετε την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τραμμένη στο πρόβλημα της διεύρυνσης και να εστιάσετε στα σημεία όπου η διαδικασία αυτή μπορεί να επιταχυνθεί. Ε, προεδρεύσατε κάτω από εξαιρετικά συνθήκες όπου ε, ήταν, ε, είχε κάνει την τάση να εστιάσει περισσότερο στη χρηματοπιστωτική κρίση και στην Ελλάδα παρά σε θέματα διεύρυνσης. Παρόλα αυτά η Ουγγαρία ανέδειξε τον ιδιαίτερο ρόλο της και την ικανότητά της να χειριστεί τα προβλήματα στην περιοχή αυτή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης τις αρετές σας και την αξία σας όσον αφορά την ε, διαδικασία προσέγγισης της Κροατίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά κάνατε πάρα πολλά και θα ήθελα να προσχωρήσω στην αρχική πρόταση του κυρίου Σβόμποντα. Ε, τι θα λέγατε αν σταματούσαμε το ρολόι και ικανοποίησαμε τις ε, προσδοκίες και τιμούσαμε το έργο το οποίο έχει γίνει. Αλλά θα ήθελα να εστιάσω παρόλα αυτά σε ορισμένα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα στην Κροατία. Η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, δεν θα πρέπει να ιδωθεί σαν ένα τρόπεο. Ε, ε, το διακύβημα εδώ είναι οι αρχές οι οποίες, και οι αξίες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από όλες τις χώρες. Όσον αφορά τις μειονότητες, η Ευρώπη έχει πολύ υψηλές προδιαγραφές. Ε, αυτό θα πρέπει να... Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνει και στην Κροατία. Και ελπίζω ότι τα πράγματα εδώ θα αλλάξουν. Συμφωνώ μαζί σας για την αξία και το γεγονός ότι η διαδικασία διεύρυνσης αφορά όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και η επιτυχία της ε, Κροατίας και στη συνέχεια του Μαυροβονίου κλπ. θα ενισχύσει τις προσδοκίες όλων αυτών των χωρών και των λαών και θα ενισχύσει την επιθυμία τους να συμβάλλουν στην σταθερότητα στην περιοχή αυτή. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Χόουιτ. Εισηγητής για τη Μακεδονία για τρία λεπτά. Ε, καταρχήν, ε, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε σήμερα. Ε, ναι, Ε, νομίζω ότι πραγματικά κάνατε ένα τεράστιο βήμα όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή. Βεβαίως θα πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες και είναι σημαντικό να συνεχίσουμε το, να στρέφουμε το ενδιαφέρον μας εδώ και να αποστέλουμε ένα μήνυμα προς όλες τις ε, χώρες ε, αυτές. Ε, υπάρχουν κάποιες ε, περιπτώσεις που εκδικάζονται στα δικαστήρια των χωρών αυτών. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ένας ε, κίνδυνος να ασχοληθούμε μόνο με τις μεγάλες χώρες, την Κροατία και την Σερβία. Εμένα με τιμά πολύ ο ρόλος μου ως εισηγητού, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στη Φιρόμ, όπου εδώ πραγματικά έχω πολλές ανησυχίες. Εδώ δεν μιλούμε για το να σταματήσουμε το ρολόι, αλλά να το βάλουμε μπροστά το ρολόι και δεν ε, και όσον αφορά τις ημερομηνίες ε, προσχώρησης για το Μαυροβούνιο και την ε, Σερβία θα πρέπει να συμπεριλάβουμε εδώ και την ΦΥΡΟΜ. Ο Επίτροπος Στέφαν Φούλε είπε την Παρασκευή ότι ελπίζει ότι θα μπορούσαν αυτό το έτος, ελπίζει ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Αναφέρθηκε στις εκλογές στην Τουρκία, έγιναν εκλογές στη ΦΥΡΟΜ ε, θα τη σχολιάσουμε. Εγώ ήμουν ε, παρόν και ε, είδαμε την έκθεση του ΑΣΕ. Η διαδικασία αυτή ήταν πετυχημένη. Θα πρέπει να αντλήσουμε βεβαίως κάποια διδάγματα αλλά θα πρέπει να χαιρετήσουμε την πετυχημένη διεξαγωγή των εκλογών στη χώρα αυτή. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περίπτωση αλλά όταν αναφέρεστε σε διμερεί θέματα τα οποία θα έπρεπε να αποτελούν τμήμα της διεύρυνσης και το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφύγει τη σύντηση αυτών των θωμάτων. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ε, κάποιες περιπτώσεις διαφόρων χωρών, τέσσερις περιπτώσεις, όπου δεν υπήρξε επιτυχία. Και η αίσθηση εκτός του Συμβουλίου ε, είναι ότι οι χώρες αυτές θέλουν να συνεχίσουν αυτές τις διμερείς συζήτησεις. Αναφερθήκατε στην Ουγγαρία λέγοντας ότι έχει ένα ε, ουσιαστικό ενδιαφέρον. Τι γίνεται με άλλες ε, χώρες που έχουν ε, ενδιαφέρον να σταματήσουν αυτές τις διμερείς συζητήσεις. Πώς μπορείτε να ασκήσετε μια επιρροή στο Συμβούλιο. κυρία Μπραντνερ για τρία λεπτά. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία που συμπερέλαβε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και θα ήθελα να χαιρετήσω το πρόγραμμα της Κροατίας για τα τελευταία χρόνια και βέβαια τους τελευταίους μήνες. Είχαμε ανησυχίε, αλλά είδαμε την ε, παρέλαση, την Gay Pride στο Split Ε, και ε, την απαγόρευσή της. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα εσφαλμένο μήνυμα από την ε, Κροατία. Δεν ξέρω πώς θα γίνουν οι μεταρρυθμίσεις τα επόμενα χρόνια σε ό,τι υπάρξει πραγματική προσχώρηση. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις και δεν θα πρέπει να αναστραφεί η παρούσα διαδικασία και θα πρέπει να εδράζεται στη διακοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ Κροατικής Βουλής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμπερίληψη της κοινωνίας των πολιτών και των ακαδημαϊκών. Και θα πρέπει η παρακολούθηση να εδράζεται στην συνθήκη. Ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αναβληθεί η βοήθεια, αλλά θα πρέπει καταρχήν να υπάρξει πολιτική πίεση, ε, περιορισμό στην χρηματοδότηση και αν σταματήσουν οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αναβληθεί η διαδικασία αλλά βεβαίως θα πρέπει να υποστηρίξουμε εκείνους τους παράγοντες στην Κροατία οι οποίοι υπερασπίζονται τις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτά όσον αφορά την Κροατία. Τώρα, όσον αφορά τις ε, διμερείς σχέσεις, την, αναφέρθηκαν εδώ οι συνάδελφοι, νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα κλειδί το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ότι αυτά τα διμερεί θέματα θα πρέπει να επιλύονται πριν από την προσχώρηση ε, σε σχέση με αυτό χάρηκα το ότι εξήρατε το διάλογο μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου αξιολογώντας τον ως θετικό και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα συνεχίσετε από την ε, πλευρά των ευρωπαϊκών χωρών και την αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου. Υπάρχει εδώ κάποια κίνηση. Ε, τι θα γίνει εάν πιέσουμε τη σερβική πλευρά το οποίο είναι ορθό. Ε, τι θα γίνει με τα δικά μας ιστορικά προβλήματα τα οποία συνεχίσουν να υφίστανται. Όπως είπε ο κύριος Φόπα, ο κύριος Βάγκελ, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι δεν ε, θα αποστείλουμε το μήνυμα ε, εντάξει για την Κροατία αλλά εδώ θα σταματήσουμε. Γιατί πολλές από τις χώρες, εγώ προέρχομαι από τη Γερμανία, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι η Κροατία δηλαδή είναι κοντά σε εμά, αλλά εδώ θα σταματήσουμε και πραγματικά θα πρέπει να αποφύγουμε κάτι τέτοιο και θα ήθελα να συγχαρώ την ε, Προεδρία η οποία συμπεριέλαβε όλη την περιοχή. Κύριος Πάσχου, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας καλωσορίσω. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ μεταφέρατε κάποιες από τις απόψεις αυτών που λαμβάνουν πραγματικά αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την διεύρυνση. Και τρίτον, μια ερώτηση. Πώς συνδυάζεται την, το καθεστώς της υποψήφιας χώρας της Τουρκίας με το ότι η χώρα αυτή γίνεται περιφερειακή δύναμη σε μια περιοχή η οποία παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον για μας. Ευχαριστώ κύριε Πάσκου. Ο κύριος Αγκουράκης. Τρία λεπτά. Μικρόφωνο κύριε Αγκουράκη. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα καταρχήν να ε, σημειώσω προς τον κύριο Υπουργό Εξωτερικών ότι παρά τις κασάνδρες που λέγανε διάφορα πράγματα εθνικιστικού χαρακτήρα και σοβινιστικού ότι δίθεν η Ουγγαρία μια μικρή χώρα δεν θα τα καταφέρει στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κατάφερε μια χαρά. Φυσικά ε, είχε την τύχη ο κύριος Υπουργό να χειριστεί και πολλά άλλα μεγάλα ζητήματα. Δυστυχώς για αυτόν είχε και τον πόλεμο στη Λιβύη, αυτή την, τον υπεριαλιστικό και την επέμβαση, τα ζητήματα της κρίσης και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αυτό που ήθελα να τονίσω κύριε Υπουργέ θα συμφωνήσω μαζί σας ενδεχομένως ότι οι παράλληλες γραμμές μπορεί να, μπορεί συναντηθούν. Η ελπίδα μου είναι όμως να μην συναντηθούν στο άπειρο, όπως γνωρίζετε, και να ζήσουμε <laughs> το σημείο της επαφής. Εννοώ δηλαδή διακαώς ε, το κόμμα μου θα ήθελε πραγματικά να λυθεί το θέμα του ονόματος με τη γειτονική χώρα, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και μια σειρά από άλλα ζητήματα, γιατί θεωρούμε πραγματικά ότι η βελτίωση των σχέσεων, οι σχέσεις καλής γειτονίας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα όχι μόνο στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Φύρομ, αλλά γενικά στα Βαλκάνια. Και από την άποψη αυτή, κύριε Υπουργέ, θα περίμενα κάτι παραπάνω και από την ε, ε, Ουγγρική Προεδρία, αλλά και από την τοποθέτησή σας, γύρω στα εξή δύο ζητήματα που μας απασχολούν πάρα πολύ. Όπως άριστα γνωρίζετε, η οικονομική κρίση του καπιταλισμού έχει χτυπήσει ιδιαίτερα σκληρά αυτή την περιοχή, γιατί ακριβώς ήταν πολύ πιο ε, πίσω, λιγότερο αναπτυγμένη. Όταν βλέπω στην Ελλάδα η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων να ζητά σήμερα την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης στη χώρα μου. Όταν γνωρίζω ότι στην Κροατία υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία που είναι αντίθετη στην ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ξέρω ότι στη Σερβία, με βάση στοιχεία του Γκάλοπ, όχι κάποιο άλλο Ινστιτούτου, κακώς αλλά έτσι είναι, οι Σέρβοι θεωρούν τον Μλάδιτς ότι δεν για, την, ε, για αυτά που προσάπτουν, τότε υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ. Ε, όπως επίσης γνωρίζετε και οι νέες χώρες που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία αντιμετωπίζουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από ότι οι παλιότερες και εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της πολιτικής της. Με αυτή την έννοια νομίζω αυτό πρέπει να πάρθει υπόψη όπως και στην περίπτωση της ε, Ισλανδίας και δυστυχώ να επιβεβαιωθεί αυτό που λέγαμε, ο φόβο μα, ότι δηλαδή η ένταξη θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Κλείνοντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τι αρχέ και το λαό τη Κροατία για τη φιλοξενία τη αντιπροσωπεία μα εκεί και να σημειώσω ότι δυστυχώ η ένταξη τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνοδεύεται με το κλείσιμο των αυπηγείων και με χιλιάδε χαμένε θέσει εργασία για του εργαζόμενου στη χώρα αυτή, χωρί να υπάρχει λύση. Η μόνη λύση που υπάρχει είναι η ανεργία και πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα είναι το μέλλον και για τι υπόλοιπε χώρε των Βαλκανίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αγκουράκη. Ο Αντιπρόεδρος κύριος Τόκες έχει το λόγο. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινώ λέγοντας ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών κύριος Μόρτη έχει γεννηθεί στο όροτα της Ρουμανίας, στην ίδια πόλη που γεννήθηκα και εγώ. Αποτελεί δηλαδή και το σύμβολο της συνεργασίας, η παρουσία του, της συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ Ρουμανίας και Ουγγαρίας. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμά που υπεστήριξε την προσχώρηση της Ρουμανίας μαζί με τη Βουλγαρία στο χώρο του Σέγγεν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ουγγαρίας. Και να σημειώσω ότι εχθές μαζί με τον Πρόεδρο Κουκάν είχα την τιμή να φιλοξενήσω την αλβανική, αντιπροσω... την αλβανική αντιπροσωπεία και να επισημάνω ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αρκετά συχνά ένα κλασικό πρόβλημα. Λόγω εσωτερικών προβλημάτων δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία τη προσχώρηση Αλβανία, δεν μπορούν να εκδώσουν κοινή δήλωση διότι η κυβέρνηση διαφωνεί με την αντιπολίτευση. Αλλά από την άλλη θα ήθελα να σημειώσω και ότι υπάρχουν ζητήματα όπου θα πρέπει τα εξωτερικά προσκόμματα να αντιμετωπίζονται. Φερρυπίν στην περίπτωση της Μακεδονίας. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι πιστεύω πως ανεξαρτήτως της διαφωνίας σχετικής με το όνομα μπορούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για προσχώρηση της Μακεδονίας. Το πιστεύω αυτό ακράδαντα και αυτή είναι η θέση την οποία προβάλλω. Και θα ήθελα εν τέλει να σημειώσω ότι τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση στην Ουγγρική Προεδρία για το έργο της. Τη συγχαίρω ο Πρωθυπουργό Βίκτορ Όλμπαν επισκέφθηκε την ε, Αλβανία στο παρελθόν. Φαντάζομαι ότι θα επισκεφθεί και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Φαίνεται δηλαδή να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις, ε, στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. παρά τις ε, επικρίσεις που έχει υποστεί και ο ίδιος και η κυβέρνησή του, εγώ θα θέλω να εκφράσω την ε, εκτίμησή μου για αυτή τη χειρονομία και τη στάση. Ξέρετε ότι είναι μια περιοχή δύσκολη εκεί και λόγω των μειονοτήτων. Ούγγροι υπάρχουν και στη Σερβία και στην Κροατία. Πιστεύω όμως ότι αντιμετωπίστηκαν κατά τρόπο ικανοποιητικό τα προβλήματα από την Ουγγρική κυβέρνηση, η οποία μπόρεσε να ρίξει γέφυρες και να αναπτύξει διάλογο με τις περιοχές. Ευχαριστώ πολύ. κύριος Λίτσεκ. Ευχαριστώ <clears throat> panie Πρόεδρε, ευχαριστώ. δεν θα χρειάζονταν τα τρία λεπτά και έτσι θα επιτρέψουμε περισσότερο χρόνο για τον ε, κύριο Υπουργό. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία για τη δουλειά της. Έργο καθόλου εύκολο θα έλεγα κατά καιρούς με το σύστημα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πτύξει, την εναλλασσόμενη δηλαδή Προεδρία, το κλειδί για την επιτυχία στις διαπραγματεύσεις, οποίες αναφερόταν ο κύριος υπουργό, είναι πάνω απ' όλα το πώς θα περάσει η σκητάλη από τη μία Προεδρία στην άλλη. Πρέπει δηλαδή να ενημερώνεται η νέα Προεδρία από την απερχόμενη για το έργο της και για την εξέλιξη των διαφορών θεμάτων. Εμείς ξέρετε Πολωνοί και Ούγγροι θεωρούμε πως είμαστε αδελφά έθνη. Ερωτώ λοιπόν κύριε Υπουργέ πώς βλέπετε τα θέματα αυτά σε σχέση με τον Πολωνό ομολογό σας. Έχετε συζητήσει τα θέματα αυτά, τι είδους εμπειρία έχετε αποκομίσει από την στάση του Πολωνού ε, Υπουργού. Ευχαριστώ. Ο τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Και εγώ από τη δική μου πλευρά ευχαριστώ θερμά για τις ε, πετυχημένες σας προσπάθειες το ζήτημα της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με την Κροατία. Η Ουγγαρία είχε πει στην αρχή ότι θέλουμε να επιδείξουμε φιλοδοξία. Το κατά πόσο ε, τηρούνται όλοι οι τύποι αυτών είναι δευτερεύων. Ε, το ζητούμενο είναι να ολοκληρωθούν. Ένα σύντομο ερώτημα. Περιμένετε κάποιες ε, ε, διαταραχές της τελευταίας στιγμής γιατί γνωρίζουμε κάποιες χώρες που ήταν επιφυλακτικές για παράδειγμα κάτω χώρες και η Σλοβενία είχε εκφράσει κάποια προβλήματα. Ε, θεωρείτε ότι θα συμβεί κάτι τελευταία στιγμή ή διαφέρονται θετικέ εξελίξεις. Όσον αφορά τη Μακεδονία, έχω, συμμερίζω με την άποψη των άλλων συναδέλφων που ε, λένε ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση με την Ελλάδα για να μην ε, μπλοκαριστεί η κίνηση των διαπραγματεύσεων. Ε, υπάρχει μια συμφωνία του 1995 όπου συμφωνήθηκε να μην μπλοκαριστεί η προσχώρηση στους διεθνείς οργανισμούς, έστω και αν δεν έχει λυθεί το θέμα του ονόματος. Νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση ξεκάθαρα με την Ελλάδα. Και ένα άλλο θέμα στο πλαίσιο αυτό. Ίσως ε, θα πρέπει να αναμένουμε εσότου αυτή κρυθεί η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο, τι θα γίνει, ποια είναι η δεδηλωμένη πρόθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Κλείνει η συζήτηση με τον κύριο Κασουλίδη. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ στην ερώτηση την οποία έκανε ο κύριος Χάουιτ για τα διμερεί προβλήματα τα οποία παρεμποδίζουν την επιθυμητή διαδικασία της διεύρυνσης. Να πω λοιπόν να ρωτήσω εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των προεδριών της θεωρεί ότι μπορεί ή πρέπει μάλλον να κάνει περισσότερα και με περισσότερη ενέργεια έτσι ώστε να βοηθήσει να επιληθούν τα διμερεί αυτά προβλήματα. Γιατί ακόμα και αν ξεκινήσει η διαδικασία διεύρυνσης, έχουμε ήδη δει και το έχουμε δει επανειλημμένα, ότι αυτά τα διμερεί προβλήματα εντάσσονται στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και τα εμπόδια αυτά τείνουν να επαναλαμβάνονται συνεχώς. σε θέματα τα οποία αφορούν άμεσα της, τη σύνδεση όπως το όνομα της συγκεκριμένης χώρας, της ΦΥΡΟΜ όπου τα Ηνωμένα Έθνη έχει κάνει, τα έχουν κάνει μια πρόθεση και στις δύο πλευρές ο Μπαν Κιμούν ο ίδιος όταν τον επισκεφθήκαμε στη Νέα Υόρκη είπε ότι η Ελλάδα είχε δεχθεί την πρόταση που έκαναν τα Ηνωμένα Έθνη και περίμεναν την απάντηση από τη ΦΥΡΟΜ μετά από τις εκλογές. Λοιπόν, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει περισσότερη ενέργεια εν πάση περιπτώσει, βοηθώντας τις δύο πλευρές να επιλύσουν το διμερές τους πρόβλημα, έτσι ώστε μια τέτοια διαδικασία διεύρυνσης να ξεκινήσει χωρίς τέτοιου είδους εμπόδια. Έχουμε δει παραδείγματα σχετικά με την Κροατία σαν παράδειγμα όπου ήρθαν στην επιφάνεια κάποια τέτοια εμπόδια αλλά αντιμετωπίστηκαν. Ευχαριστώ κύριε Κασουλίδη. Θα δώσουμε τώρα την δυνατότητα στον Υπουργό. Λοιπόν κύριε Υπουργέ έχετε τον χρόνο που είναι απαραίτητος μιας και ξεκινήσαμε με μια κάποια καθυστέρηση ε, για να απαντήσετε σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τα σχόλια αλλά και τις παρατηρήσεις. Θα προσπαθήσω να είμαι τουλάχιστον συντομότερος από ό,τι ήμουν στις αρχικές μου παρατηρήσεις. Ζητώντας συγγνώμη που με τόσο. Αν και θα Πρέπει να επισημάνω ότι είχα και άλλα θέματα υπόψη, τα οποία δεν εξέθεσα. Χάρη σε ερωτήσεις ε, μπορώ τουλάχιστον να απαντήσω τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα, ώστε να τον πιο σύντομο. το ενδιαφέρον που μπορεί να τρέφει η Ουγγαρία για τη διεύρυνση. Και ολόκληρης βέβαια της ε, ζώνη Βαλκανική, τη Δυτική ε, βαλκανική είναι σαφέ. Το έχουμε επισημάνει σε πολλέ συνεδριάσει, συναντήσεις, συνομιλίε. Και αυτό νομίζω παρουσιάζεται κατά τον καλύτερο τρόπο και από τον Αντιπρόεδρο Τουρκές με την επισήμανση ότι ο Πρωθυπουργό ήταν στο Βελιγράδι, μετά στο Μαυροβούνιο, στο, στις διάφορες χώρες της και εγώ ίδιος ε, έχω τακτικά συναντήσεις με τους υπουργούς των εξωτερικών ε, της ε, περιοχής. Φυσικά και μας ενδιαφέρει και δεν αποκρύπτουμε άλλο στο γεγονός ότι έχουμε και συμφέρον εθνικό στη σταθερότητα και την ευημερία και την ευρωπαϊκή προοπτική των κρατών αυτών. Δεν αναφέρθηκα εκτενώς στις προκλήσεις, υπάρχουν προκλήσεις σε ορισμένες από τις χώρες αυτές. Βλέπουμε κάποια ακτίδα ελπίδας για τη Βοσνία, όντως, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις προσπάθειες της, ε, ε, της εκπροσώπου της Καθιάς, η οποία έπεισε να μην γίνει το δημοψήφισμα που είχε προβλεφθεί τουλάχιστον μην γίνει αμέσω να αναβληθεί, άρα έχει κάπως διευκολύνει την κατάσταση. Πάντως επισημαίνω ότι συμφέρον όλων μας είναι τόσο στη Βοσνία όπως και στην Αλβανία, σε τέτοιου χώρες, να προχωρήσουν τα πράγματα κατά τρόπο θετικό. Το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών πρέπει να επισημάνω έχει στο θέμα, στην ημερήσια του διάταξη το θέμα της Αλβανίας τη Δευτέρα 20 Ιουνίου. Και θα διατυπώσουμε και τα σχετικά συμπεράσματα εμείς. Θα δείτε το κείμενο. Το κύριο ε, μήνυμα θα είναι ένα, μια φιλική προειδοποίηση να αλλάξουν στάσεις ε, σε εξέλιξη που παρατηρούμε τώρα. Για το Διεθνές Δικαστήριο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ε, διαδικασίες, όχι μόνο σχέση με το αλλά και γιατί περιμένουμε να αντιδράσουν και τα εθνικά δικαστήρια. Χτες συζήτησα με τον κύριο Μπάμερτς ε, σε μια συνάντηση ε, εκτενώς για τα θέματα αυτά και συμφωνούμε ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί. για τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινούν οι διαδικασίες. Εγώ ως Ούγκρος ε, εθνικά δηλαδή μιλώντας μπορώ να πω ότι ναι συμφωνώ και θα πρέπει να γίνει σχετική σύσταση προς την Επιτροπή. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε και να αρνηθούμε ως Ευρωπαίοι ότι χρειάζεται η συμφωνία των ε, ευρωπαϊκών κρατών μελών στο σύνολό τους και εδώ θα ήθελα να επεκταθώ λίγο περισσότερο, γιατί έχουμε να κάνουμε λεπτά ζητήματα, ευαίσθητα ζητήματα, γιατί αφενός με, γνωρίζουμε ότι όλοι θέλουμε να δώσουμε μια χειρά θέλουμε να υποστηρίξουμε την υπόθεση αυτή, να ενθαρρύνουμε. Να αποστείλουμε και μήνυμα ότι θα ήταν προτιμότερο να προχωρήσουν οι χώρες στη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να προκύψει εξή ή άλλη συνέπεια. Αλλά την συμφωνία. Δεν μπορούμε να τη συνάψουμε εμείς. Εάν δεν το θέλουν οι χώρες, δεν μπορεί κανείς έξωθεν να τους επιβάλλει μία συμφωνία. Σε ορισμένε περιπτώσεις βέβαια καταφέρνουμε να φτάσουμε σε επιτυχία. Η Κροατία φέρει Η προσχώρηση Κροατίας θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς μια συμφωνία διαιτησίας με τη Σλοβενία. Έγινε όμως. Και θα εγκρίνει το Σλοβενικό Κοινοβούλιο, ελπίζουμε, το κλείσιμο των διαπραγματεύσεων την προσεχή Παρασκευή. Άρα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Από την άλλη όμως πρέπει να είμαστε και Θα πρέπει να δούμε ότι όταν προκύπτουν διμερεί ζητήματα έχουμε κάποιο ρόλο να διαδραματίσουμε με ένα, αλλά πρέπει να τον διαδραματίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή, σύνεση και σεβασμό των εξουσιών των εν κρατών. Για την Τουρκία συμφωνώ μαζί σας απολύτως και εγώ ε, συμμερίζομαι τα συγχαρητήρια, γι' αυτό και αναφέρθηκα στη δήλωση Μπαρόσο και Ρομπόη. Συμμερίζομαι ως προς το περιεχόμενο και την ουσία της δηλώσης αυτές. Ε, πιστεύω ότι απεστάλλει και το κατάλληλο μήνυμα πλέον για το Gay Pride. Κυρία Πρατνάρ. Νομίζω ότι αποτελεί απόδειξη ικανοποιητική πως πρέπει να επιτευχθεί μία πρόοδος περαιτέρω. Παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή βέβαια και για την ε, Κροατία. Υπάρχουν ε, ζητήματα νομοτεχνικά, νομικά που πρέπει να διευκρινιστούν. Θα πρέπει να δούμε πώς θα τα χειριστούμε. Ο κύριος που κάθεται δίπλα μου θα μπορούσε να σας δώσει περισσότερες απαντήσεις για την υπόθεση αυτή. Πάντως εγώ προσωπικώς μπορώ να πω ότι τρέφουμε αισιοδοξία. Είμαστε αισιόδοξοι. Και βέβαια, παρεμπιπτόντως θα αναφέρω ότι το κλειδί για την επιτυχία μια διεύρυνση είναι στα εθνικά κοινοβούλια, γιατί αυτά καλούνται να κυρώσουν την διαδικασία της διεύρυνσης για την κάθε χώρα. Ίσως είναι τυπικό αυτό θα μου πείτε, αλλά πάντως υπάρχει. Και το θέμα πιστεύω θα επιληθεί κατά τρόπον ικανοποιητικό για όλους. Η αναγνώριση του κοσφοπεδίου. Ξέρουμε ότι είναι διχασμένα τα κράτη-μέλη. Μπορούμε να το συστήσουμε σε φιλική βάση αν θέλετε αυτοί που αναγνωρίζουν με αυτού που δεν αναγνωρίζουν το κοσμοπέδιο μπορούμε να το συζητήσουμε και το πράττουμε του, σε, σε κάθε συζήτηση φιλική, άτυπη με του φίλου. Η ε, μεν και η δε το συζητούμε. Γνωρίζουμε η μεν τα επιχειρήματα των δε. Προσπαθούμε να πείσουμε, εγώ δηλαδή από πλευρά μου προσπαθώ να πείσω εκείνου που δεν αναγνωρίζουν το κοσμοπέδιο, αλλά γνωρίζουμε βέβαια και τα όρια. Ε, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι τέτοιο έξωθεν και πάντως ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω. Και γι' αυτό και υποστηρίζουμε το διάλογο μεταξύ της Πρίστινα και του Βελιγραδίου, τους πέντε γύρους που αποτέλεσαν ευκαιρία όχι μόνο για πολύ ορθολογικό διάλογο, αλλά και για ουσιαστική πρόοδο σε κάποια στο περιορισμένα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν, τεχνικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν, χωρίς να κρυθεί το ζήτημα του καθεστώτος. Τουρκία. Εγώ δεν βλέπω εδώ αντίφαση μεταξύ της προοπτικής για ένταξη της Τουρκίας και της ανάπτυξης ε, της παρουσίας Τουρκίας στην περιφερειά της ως μεγάλης δύναμης περιφερειακής. Θα έλεγα μάλιστα ότι μέχρι του έρθει η ώρα για την προσχώρηση της Τουρκίας θα έχει ακόμη ενισχύσει την παρουσία της ως ε, περιφερειακής δύναμης αλλά αυτό σημαίνει και την δύναμη που θα αποκτήσει η Ευρώπη ταυτόχρονα. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Θέλουμε αυτή η μεγάλη περιφερειακή δύναμη την Τουρκία μέσα στην Ευρώπη ή εκτός αυτής. Αυτό είναι ένας, ένα ζήτημα στρατηγικό, μια επιλογή θεμελιώδης που θα πρέπει να αναλύσουμε και εμείς έχοντας πράξει αυτή την ανάλυση, έχουμε προχωρήσει αυτή την ανάλυση, καταλήγουμε ότι θέλουμε τη μεγάλη αυτή περιφερειακή δύναμη να την έχουμε μέσα στην Ευρώπη. Κάποιοι άλλοι μπορούν να καταλήγουν σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει όμως προτείνουμε τώρα προχωρούμε, να προχωρούμε τώρα σιγά σιγά στις διαπραγματεύσεις αντιμετωπίζοντας ε, προβλήματα όχι μόνο από πλευράς μας αλλά και από πλευράς των Τούρκων και αναφέρομαι εδώ σε συμπληρωματικό πρωτόκολλο ε, και, να, και θέλω να επισημάνω επίση ότι είναι προ το συμφέρον τη Ευρώπη να έχει μέλο τη στην Τουρκία, τουλάχιστον κατ' εμά. Ένα άλλο ζήτημα Δεν θέλω να επισημάνω για την Ουγγαρία συγκεκριμένα ότι να είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 7 χρόνια. Η εμπειρία μας είναι εν γέννη θετική. Η χώρα μου έχει αποκομίσει πολλά ωφέλη βέβαια από την ε, προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το αρνούμαστε. Προβλήματα επίσης είχαμε, οικονομικά και άλλα, τα οποία όμως δεν τα αποδίδουμε στην προσχώρηση. Είναι δικά μας σφάλματα. Είναι λάθη δικά μας. Όπω είπα δηλαδή και για να είναι απόλυτα σαφέ, έχουμε ωφεληθεί πάνω απ' όλα από την προσχώρησή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφέ ότι έχουμε όφελο. Γι' αυτό και είμαστε πεπισμένοι ότι τα κράτη που θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέλλον η Κροατία πρώτα και τα υπόλοιπα μετά, θα ωφεληθούν πάνω απ' όλα από την ε, προσχώρηση. Η συνεργασία με την Πολωνία έχει προχωρήσει πολύ καλά. Θα συνεχίσει ασφαλώς και με το, επόμενη τρία Ανδρία με το επόμενο τρίο που θα αναλάβει με πρώτη την Πολωνία. Είναι ένα κεντροευρωπαϊκό έτος το φετινό, με την Ουγγαρία πρώτη και την Πολωνία δεύτερη στην Προεδρία. Και είναι ενδιαφέρον ότι νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κεντρικής Ευρώπης κιόλας, μπορούν ε, να έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι μπορούν να διοικήσουν αποτελεσματικά στο εξάμεινο την Προεδρία τους εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ιδιαίτερα σημαντικό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα περισσότερα ζητήματα, γιατί σήμερα συστήσαμε εδώ την διεύρυνση, αλλά και σε άλλα θέματα, στην πολιτική της συνοχή, στη γεωργική, την ενεργειακή πολιτική. Ε, σε πολλά από τα θέματα, λοιπόν, στα περισσότερα, ένα από τα συμπεράσματα που μπορεί κανείς να διατυπώσει, να αποκομίσει από αυτήν ε, περίοδο του εξαμήνου μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δούλεψε. Δούλεψε και δούλεψε κυρίως στον τομέα της διεύρυνσης. Γιατί ήταν σαφές το μήνυμα από πλευράς μας και αυτό το λέω εκ μέρου των λεγόμενων νέων μελών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής των κρατών της Ευρωπαϊκής Ευρώπης. Δουλέψαμε, δώσαμε το μήνυμα ότι θέλουμε τη διεύρυνση. Και νομίζω διαδραματίστηκε αυτό το ρόλο του. Προβλήματα τη τελευταία στιγμή δεν αναμένω και θα ήθελα να καθίσω σαφέ με μια δήλωση ότι δεν αναμένω τέτοια προβλήματα. Και αν ήθελα να μην είμαι τόσο σοβαρό, ε, θα έλεγα ότι αν δεν περίμενα τέτοια προβλήματα, δεν θα έλεγα ότι δεν περιμένω προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει όμω, για να παραμείνω σοβαρό, ε, υπογραμμίζω ότι δεν αναμένω ε, προβλήματα τη τελευταία στιγμή. Για την ε, διακυβερνητική και τη διαδικασία που ξεκίνησε σε σχέση με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πιστεύουμε ότι θα, βρούμε μια, θα δούμε μια εξέλιξη κάπου τον Οκτώβριο και αναλόγως τις πολιτικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Άλλο ένα πράγμα που αναφέρθηκε βέβαια δεν είναι ακριβώς αντικείμενο των σημερινών μας συνομιλιών αλλά ακούστηκε, έγινε λόγος για το Σέγγεν και αυτό είναι πολύ σημαντικό η Προεδρία μας ακολούθησε μια πολύ βασική αρχή και θα ήθελα να την υπογραμμίσω, να την περιγράψω πολύ πολιτική περιεκτική. Τι σημαίνει περιεκτικότητα. Πάνω απ' όλα σημαίνει διεύρυνση. Έχουμε συζητήσει τη διεύρυνση, την, τα, είπαμε τώρα, ξέρουμε τι έχει επιτευχθεί, πού αποσκοπούμε για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα προσεχή χρόνια. Περιεκτικότητα όμως σημαίνει και την περίληψη της ε, Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο του Σέγγεν. Και εμείς από πλευρά μας κάναμε ό,τι μπορούσαμε για το στόχο αυτό. Πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε ε, να αναζημιώσουμε ότι υπάρχει μια, κάποια επιτυχία, κυρίως σε σχέση με την κατάσταση που παρουσίασαν πριν από δύο-τρει μήνες. Και επίσης, γιατί πρέπει να ληφθεί και απόφαση, ε, συμπερίληψη σημαίνει, συμπερίληψη σημαίνει ε, και συμπερίληψη στις κοινωνίες διάφορων τμήματων αυτών των κοινωνιών, όπως φερειπίν τον Ρωμά. Εδώ πάλι έχουμε την περιεκτικότητα ως πολιτική και πιστεύω ότι και αυτό αποτέλεσε ε, λίθο θεμέλιο της Προεδρίας μας. Που προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην πολιτική μας και για τη διεύρυνση. Αυτά λοιπόν είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή, για τη συνεργασία, για την υποστήριξη που προσφέρατε στην Ουγγρική Προεδρία σε αυτούς τους πεντέμισι μήνες. Τελευταία στη ε, παρατήρηση και ελπίδα να μην σταματήσουν τα ρολόγια, να συνεχίσει ο χρόνος να τρέχει. Ούτως ή άλλως το χρόνο δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Και αν αντιληφθούμε τι απαιτούν οι καιροί, αυτοί οι μεταβαλλόμενοι καιροί, οι εποχές αυτές, και αν δούμε ευρύτερα τι συμβαίνουν παράλληλα, ευρωζώνη, κρίση, παγκόσμιες απειλές, είναι βέβαιο ότι δεν έχουμε περιθώριο να επιβραδύνουμε τους, ρυθμού τους ρυθμούς μας. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τους δείκτες του ρολογιού. Πρέπει να προχωρήσουμε, να ολοκληρώσουμε και να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνατε αυτούς τους έξι μήνες, σας ευχαριστώ για την προσοχή που στρέψατε στο Κοινοβούλιο και πράγματι ελπίζω να μοιρασόμαστε όλοι την επιθυμία να συνεχίσουμε τις προσπάθειες έτσι ώστε να πετύχουμε και τους άλλους κοινούς στόχους. Ευχαριστώ λοιπόν και καλή συνέχεια. Σας χαιρετώ κύριε Υπουργέ λοιπόν. Θα σας χαιρετήσω και εγώ. Αφήνω την Προεδρία στον συνάδελφο Πάσκου, ο οποίος θα συνεχίσει με την ημερήσια διάταξη. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας. Αγαπητοί φίλοι, ας συνεχίσουμε, γιατί έχουμε μια φορτωμένη ημερήσια διάταξη και θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε όλα τα σημεία που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Για την αρχή ε, θα δώσω το λόγο στο πρόεδρο του Κοινοβουλίου για να... Θα δώσω στο, στον κύριο για να μας μιλήσει για το θέμα των ανθρωπιστικών καταστροφών. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ανακοίνωση της Επιτροπής για το 2010 προς μια πιο ισχυρή απόκριση στις ανθρωπιστικές καταστραφές. Ο ρόλος της ανθρωπιστικής συνδρομής καταδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω βελτίωση, ε, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, συνεκτικότητα και ορατότητα της Ευρωπαϊκής Συνδρομής στο σύνολό της. Επίσης, δηλώνει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να συμπεριλαμβάνει πρόληψη, επαρκή προετοιμασία και απόκριση σαν την πιο αποτελεσματική στρατηγική για βελτίωση. Ε, ε, διατηρώντας όλα αυτά τα ευρήματα κατά νου και σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης σαν μία από τις θεμελιώδεις ιδρυτικές αρχές στην Ευρώπη, κατά, στη γνωμοδότησή μου εστιάζω στην ανάγκη για, μια, για έναν καλύτερο συντονισμό για μια πιο ισχυρή και πιο συνεκτική δυνατότητα απόκρισης ενισχύοντας τα επιμέρους εργαλεία. Η συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει νέες νομικές βάσεις και με τον τρόπο αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες συντονισμού. Η δημιουργία της εξωτερικής υπηρεσίας παρέχει τη δυνατότητα να συντονίσουμε και να βελτιώσουμε τη συνεκτικότητα μεταξύ απόκρισης της καταστροφές και, τις, και στοιχεία που σχετίζονται με την πολιτική ασφαλείας. Μεγαλύτερος πολιτικός συντονισμός ε, απαιτείται ε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, εξωτερικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την ΚΕΠΑ, καθώς και των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της γνωμοδότησης είναι η χρήση των στρατιωτικών μέσων σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες ε, γραμμές του Όσλο και σαν έσχατο μέσο μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ε, απόκριση στις, ε, την αντίδραση στις καταστροφές. Επίσης τονίζω την ανάγκη για μια πιο περιεκτική στρατηγική επικοινωνίας ούτως ώστε να αυξηθεί η ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ευεργετούμενες χώρες και για μια καλύτερη κατανόηση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τόκες. βλέπετε πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σημαντικό θέμα. Ο κύριος ε, Ντόκες ε, επεσήμανε τα σημαντικότερα σημεία αυτής της προβληματικής. Ο κύριος και ο ηγητής, έχει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κρίνω θετικά την πρόταση. Συγκεντρώνει κάποιες ιδέες τις οποίες η Επιτροπή μας έχει επαναλάβει στο παρελθόν, ιδιαίτερα στην έκθεση Αλμπερτίνη για την ΚΕΠΑ. Όχι και την ανάγκη να ενισχυθεί η σύγκληση και η συνοχή ανάμεσα στα μέσα που έχει η ε, εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα διαχείρισης κρίσεων. Οφείλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε κυρίως γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος μπροστά μας, ένας κίνδυνος μιας κάποιας μιας κάποιας δυσκολίας στο να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την κοινοτική διάσταση βοήθειας ανθρωπιστικής και την δυνατότητα διαχείρισης κρίσης που έχουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για διαφορετικά μέσα με διαφορετικούς στόχους, αλλά στην καθημερινή, αν θέλετε, ζωή, οι κρίσεις αυτές πάρα πολύ συχνά είναι κρίσεις όπου οι φυσικές καταστροφές, οι ανθρώπινες πλευρές συνδέονται, συνδυάζονται και οδηγούν στην ανθρωπιστική βοήθεια. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει βέβαια να κρατήσει την αυτονομία της, αλλά από την άλλη να δώσει κάποιες δυνατότητες πολιτικής παρέμβασης που θα καταστήσει την ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεσματικότερη. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί η διάσταση αυτή η οποία όπως είπα μερικές φορές δεν συνδυάζεται με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτό είναι το πνεύμα της γνωμοδότησης, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Και εδώ έρχεται και η παρατήρηση της δυνατότητας χρήσης στρατιωτικών δυνατοτήτων για τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Κάτι τέτοιο είχε γίνει και στο Πακιστάν, όπου ε, ακριβώς στο όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συντονίστηκε η χρήση των αεροπορικών μέσων από στρατιωτικές υπηρεσίες. Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να εντάσσονται ή μάλλον θα πρέπει να σέβονται τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων μέσων και οργάνων που έχει στη διάθεσή της η Ένωση. Υπάρχει ένας επίτροπος για την ανθρωπιστική βοήθεια και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να αμφισβητηθεί αλλά από την άλλη σε λειτουργικό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί η συνέργεια και η συνοχή. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι το πνεύμα της συγκεκριμένης γνωμοδότησης Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες, κάποιες από αυτές μπορούν να βελτιώσουν την πρόταση, η τροπολογία της Μπρέντνερ σαν παράδειγμα, αλλά γενικά είναι ένα κείμενο που μπορούμε να δεχτούμε εύκολα. Ευχαριστώ κύριε Γκουαλτιέρη, κυρία Μπρέντνερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της έκθεσής σας και νομίζω ότι είναι σημαντική η έκθεση γιατί κάθε φορά υπάρχει κάποια καταστροφή ε, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα, έστω και αν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια καταστροφή. Είναι σημαντικό να οικοδομήσουμε το δυναμικό της απόκρισης. Θα ε, έγινε αναφορά στην ανάγκη συνοχής και συντονισμού αλλά δεν είμαι ακόμα απολύτως βέβαιη ε, σε σχέση με τη διάκριση των ρόλων μεταξύ εξωτερικής υπηρεσίας ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για, για την ανθρωπιστική βοήθεια. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι αναγκαίο να κινητοποιηθεί όλο το πλωστάσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και νομίζω ότι είναι αναγκαίο να τηρηθεί ουδετερότητα όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν θα πρέπει δηλαδή να την αναμειγνύουμε με πολιτικούς στόχους και είναι σημαντικό να κρατήσουμε τις ε, ε, δομές αυτού του θεσμικού οργάνου ξεκάθαρα διακριτές από πολιτικές ιδέες. Ε, θα πρέπει λοιπόν να είναι ανεξάρτητη και ουδέτερη πολιτικά η ανθρωπιστική βοήθεια διότι ακριβώς ε, ο στόχος είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και όχι η επίτευξη πολιτικών στόχων. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι επιτόπου ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις τους κλπ. κλπ παιδιά που θέλουν να σωθούν, και λοιπά, να σωθούν κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η ανεξαρτησία και η ουδετερότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικέ. Κάτι το οποίο δεν σημαίνει ότι σε ορισμένε περιπτώσει, έστω και σε πολλέ περιπτώσει, δεν χρειάζεται μία συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Δεν θα ήθελα να το αποκλείσω εν γέννη, αλλά νομίζω ότι βασική αρχή θα πρέπει να εγγυάται την ουδετερότητα της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεύτερον, επειδή δεν μιλούμε μόνο για το ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να πράξουν και χώρες μέλη, νομίζω ότι πράγματι είναι ένα θέμα ελληνική, αλλά και ευθύνη. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι χώρες μέλη έχουν ακόμα τις δυνατότητες ή μπορούν να οικοδομήσουν τις δυνατότητες που είναι αναγκαίες για την ανταπόκριση στις κρίσεις. Ε, ε, δεν θα πρέπει να υπάρξει μια, ένας, ένας ανταγωνισμός μεταξύ των... Ε, όχι, συγγνώμη, δεν θα πρέπει να υπάρξει ανάληψη αυτής της αρμοδιότητας από ορισμένε χώρες που έχουν περισσότερα χρήματα, αλλά θα πρέπει να αναλυφθεί η ευθύνη από όλε τις χώρες ε, ξίσου. Ε, αυτό λέω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 11. Σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι στο ανθρωπιστικό πεδίο τα βασικά συντονιστικά όργανα, το βασικό συντονιστικό όργανο είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Και ε, πολλές χώρες και εκτός της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, εκεί είναι το βασικό συντονιστικό όργανο. Αυτό είναι το βασικό συντονιστικό όργανο και θεωρώ ότι έστω και αν υπάρχει βελτίωση του συντονισμού θα πρέπει να ενταχθεί στον μηχανισμό των Ηνωμένων Εθνών γιατί αυτός είναι ο βασικός παράγων. Κατά τα άλλα πραγματικά υποστηρίζουμε τα περισσότερα, το μεγαλύτερο κομμάτι της έκθεσης. Ευχαριστούμε πολύ ο Hans Das εκ μέρους της Επιτροπής είναι υπεύθυνο για την ε, κατεπηγούσα απόκριση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης και θα ήθελα να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου σε αυτή την Επιτροπή για τη σημασία που προσδίδει σε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου για να πιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένα ζητήματα θεσμικής φύσεως. Για παράδειγμα, το ρόλο της ΥΠΑ της εκπροσώπου στο πάνω σχέδιο και θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα θεσμικά ζητήματα. Η πολιτική προστασία και η ανθρωπιστική βοήθεια καταρχήν είναι τα βασικά εργαλεία μέσω των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται στις καταστροφές. Δεύτερον, η πολιτική προστασία και η ανθρωπιστική βοήθεια και οι δύο συμπεριλαμβάνουν συνδρομή για τη διάσωση ανθρώπινων ζώων. Συνεπώς θα πρέπει να παρέχονται αμέσως μετά τις καταστροφές. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο χρόνος είναι πολύ ουσιώδης όσον αφορά την προστασία και την παροχή ανθρωπιστική βοήθειας, οι οποίες θα πρέπει να παράσχονται τάχιστα. Κάθε, μετρό λεπτά, ε, κάθε λεπτό μετράει και η Επιτροπή ανησυχεί ως, ε, για την δημιουργία ανησυχεί για τη δημιουργία άλλων ε, οργάνων συντονισμού. Το σύνολο του μηχανισμού συστάθηκε για να διευκολύνει την συνεργασία μεταξύ χωρών μελών και την απόκριση της καταστροφές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, αποφασίστηκε ότι ο μηχανισμός αυτός μπορεί να διατεθεί και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνήθηκαν συγκεκριμένοι κανόνες συντονισμού με τις χώρες μέλη. Επόμενο σημείο. Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εκτός από την ΚΕΠΑ. Και ε, αυτό είναι το θέμα. Αυτή, αυτό ισχύει και για την ε, πολιτική προστασία και την ευρωπαϊκή βοήθεια όπου υπάρχει μια νομική προστασία στη συνθήκη και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία είναι υπεύθυνη η Επιτροπή. Και όταν λοιπόν υπάρχει δράση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό μπορεί να διδευθεί με νομικούς όρους σαν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία των Πολιτών. Η χρήση του όρου συντονισμό στο πλαίσιο αυτό, γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι προβληματική. Το πρόβλημα είναι ότι ο όρος συντονισμός μπορεί να καλύπτει να έχει πολλές διαφορετικές έννοιες και κάποιες αμφισημίες. Για ορισμένους σημαίνει έλεγχος και καθοδήγηση για άλλους ανταλλαγή πληροφοριών. Στην ε, ε, ανταπόκριση στις καταστροφές ε, περισσότερο αναγκαία είναι η σαφήνεια εν σχέση με το ποιος κάνει τι και ποιος είναι υπεύθυνο για αυτή. Γι' αυτό υποδεικνύουμε να μένουμε στην γλώσσα της συνθήκης και να μιλούμε περισσότερο για συνεκτικότητα και συνοχή της ευρωπαϊκής δράσης και να μην αναφερόμαστε σε ζητήματα συντονισμού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Επιτροπή και εντός της Επιτροπής, ε, ιδιαίτερα η Επιτροπής Γεωργίευα, είναι η πρώτη υπεύθυνη για καταστροφές στο ευρωπαϊκό επίπεδο, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είμαστε κάπως σαν ε, στεντοφόρα στην περίπτωση αυτή που καλούμαθα να συνδράμουμε ανθρωπιστικά χωρίς καθυστερήσεις. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη, θα πρέπει να είναι ουδέτερη και θα πρέπει επίσης να σέβεται τις βασικές αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας εν γέννη. Θα πρέπει να έχει πολιτικό χαρακτήρα. Βεβαίω, παρέχοντας αυτή τη συνδρομή συνεργαζόμαστε στενά με άλλους γιατί καμία καταστροφή δεν μοιάζει με την άλλη και θα πρέπει να εξασφαλίσετε η συνοχή και υπό την έννοια αυτή ε, συνεργαζόμαθα πάντοτε στενά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και εξασφαλίζουμε μια συνοχή στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Δράσης. Αλλά η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την πρώτη απόκριση στις φυσικές καταστροφές και ε, σε αυτό αναφέρεται η ανακοίνωση αυτή. Ε, η, Επιτροπή, η πολιτική διάσταση των πολιτικών κρίσεων που είναι η διάσταση Β αφορά ε, βεβαίως περισσότερο την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Εν κατακλείδη απομένει αρκετή δουλειά να γίνει θα υπάρξουν διευθετήσει ε, μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά κατά την άποψή μου δεν χρειάζονται άλλα επίπεδα συντονισμού που ενδεχομένω θα δημιουργήσουν επικαλύψεις και θα μειώσουν την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα της ανταπόκρισης στις καταστροφέ. Η συνοχή θα πρέπει να επιτευχθεί ε, μέσω σωστής επικοινωνίας, σωστής ανταλλαγής πληροφοριών και πρακτικής συνεργασίας. Θα ήμουν ευγνώμων προς την εισηγήτρια και τα μέλη της Επιτροπής εάν τα θέματα αυτά έβρισκαν μια σωστή διατύπωση ιδιαίτερα στην πρώτη παράγραφο της έκθεσης. Ευχαριστώ. Είμαι πεπισμένος ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος και πολλά από τα θέματα αυτά θα λυθούν υπόψη εκεί που πρέπει. Η γνώμη μου είναι ότι οφείλουμε να λάβουμε, όψη, να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα γιατί νομίζω ότι αυτά τα θέματα είναι πολύ πιο σημαντικά από οποιουσδήποτε αδικαιολόγητους ανταγωνισμούς και ζήλες ανάμεσα στα όργανα. Πρέπει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια λοιπόν και είμαι σίγουρος ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί. Η επόμενη συζήτηση για το θέμα θα γίνει στις 21 του μηνός. Η ψηφοφορία θα γίνει τον Ιούλιο στην αρμόδια επιτροπή και το ίδιο θα συμβεί και με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του Προέδρου Παντσέρη Πρόεδρου της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ που μόλις επισκέφθηκε το Μαγκρόπο. Βλέπω μαζί του και την κυρία Μπουάιντα που είναι η ομόλογός του ε, από πλευράς Μαρόκου. Και οι δύο νομίζω θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλά το τι συμβαίνει. Αντώνιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Volevo solo fare un piccolo report di questa θα ήθελα να σας μεταφέρω μια έκθεση σύντομη της συνάντησης που οργανώθηκε στο Μαρόκο από τις 16 μέχρι τις 20 Μαΐου στο Ραμπάτ, στο Αγιούν και στην Καζαμπλάνκα. Υπάρχουν αρκετά σημαντικά θέματα όπως οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις, η αποκέντρωση, τα θέματα τα μεταναστευτικά, τα οποία ξέρετε ότι υπάρχουν και επιμέρους θέματα που αφορούν την αλληλεία και τη γεωργία. Γι' αυτό το τελευταίο θέμα συζητήσαμε με τον Μαροκινό Υπουργό Γεωργίας, ήταν σημαντική η συνάντηση, όχι μόνο γιατί μας βοήθησε να καταλάβουμε τα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή χαίνουν, αλλά και να ακούσουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα αυτά. Προσκάλεσε ο Υπουργό άλλωστε του Μαρόκου την Επιτροπή Γεωργίας και την Επιτροπή Αλληλείας να πάνε στο Μαρόκο για να δούνε πράγματι πού βρίσκεται το επίπεδο εφαρμογής της πολιτικής αυτής ε, και στις δύο πλευρές και στους δύο τομείς μάλλον. Εγώ έστειλα μια επιστολή και στην πρόεδρο της Επιτροπής Αλίας, την κυρία Φράγα Εστέβες, έτσι ώστε να λάβει υπόψη της αυτή την πρόσκληση και να μπορέσει το ταχύτερο δυνατόν να την πραγματοποιήσει. Συναντήσαμε επίσης και τον Υπουργό Εξωτερικών Φασά Φαρή, Και εκεί η συζήτηση ήταν σημαντική, πολύ χρήσιμη για μας. Εκφράστηκε η διάθεση του Υπουργού να προσκαλέσει την Μικτή Επιτροπή στο επόμενο Συμβούλιο Σύνδεσης που θα διεξαχθεί το Δεκέμβριο. Θα στείλουμε μια κοινή επιστολή με την κυρία Μπουντάια και προς τον Επίτροπο Φίλε έτσι ώστε να περάσει από τα λόγια στις πράξεις γιατί εφόσον έχουν υπάρξει εξελίξεις είναι σαφές ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει την Επιτροπή τη διακοινοβουλευτική. Κατά τη διάρκεια των εργασιών έγινε δεκτή και μία πρόταση για την αποκέντρωση ή περιφερικοποίηση στο Μαρόκο, ένα ψήφισμα ε, καταδίκης των τρομοκρατικών ε, ενεργειών που έγιναν στο Μαρακές πρόσφατα και προετοιμάζουμε και άλλα δύο σημαντικά έγγραφα τα οποία επεξεργαζόμαστε. Το ένα αφορά την ε, πολιτική της μετανάστευσης και το άλλο την πολιτική της ανάπτυξης στα πλαίσια της νέας πολιτικής γειτονίας. Κάναμε μια συζήτηση σε βάθος όλων αυτών των προβλημάτων που είχε σαν στόχο να εμφαρίνει τη δημιουργία, την εμβάθυνση μάλλον των πολιτικών μεταρρυθμίσεων και τον Ιούλιο θα υπάρξει και ένα δημοψήφισμα στο Μαρόκο για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και θα υπάρξουν και πρόορες εκλογές τον Οκτώβριο, δύο σημαντικές χρονικές στιγμές δηλαδή. Τέθηκε το θέμα της αποκέντρωσης των εξουσιών, το θέμα της αποκέντρωσης στον τομέα της ε, οικονομίας τέθηκε σε συζήτηση και αυτό το οποίο είπε η αυτομεγαλειώτης για τις μεταρρυθμίσεις και για την συνέχιση της δυνατότητας διορισμού του Πρωθυπουργού πάντα από τον Βασιλέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί. Εμείς επιμείναμε στις αλλαγές που είναι απαραίτητες στον τομέα της ελευθερίας του τύπου διεκδικήσαμε ένα ισχυρότερο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, κάναμε συναντήσεις και στην Καζαμπλάνκα και στο Ελαγιούν με νέους πανεπιστημιακούς, φοιτητές μάλλον από το Πανεπιστήμιο και ζητήσαμε να υπάρξει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα από όλους για το θέμα της Δυτικής Σαχάρας Είχαμε επίσης και συνάντηση με την αντιπροσωπεία της Ένωσης του Αγιούν. Μας ε, υπόθηκε ότι η κατάσταση ήταν σχετικά σταθεροποιημένη και στα πλαίσια της λειτουργίας της Τριμερούς Επιτροπής για τον έλεγχο σεβασμού κατάψασης, κατάπαυσης του πυρός Υπάρχουν κάποια θέματα που μένει όμως να αντιμετωπιστούν. Το θέμα της απογραφής του πληθυσμού είναι ένα από αυτά και αυτό είναι αντικείμενο δημοψηφίσματος. Το δεύτερο το οποίο δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε ε, είναι ο προβληματικός ρόλος του τύπου ο οποίος λειτουργεί προπαγανδιστικά και δεν βοηθά την διαδικασία αυτή. Αυτά μας είπε ο εκπρόσωπος, ο υπεύθυνο της αποστολής Μίνου, στην οποία συμμετέχει ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει εμείς και στη δική μας συνάντηση και στα πλαίσια της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και μετά από συναντήσεις που είχαμε με εμπλεκομένους είπαμε ότι ο υπεύθυνο της αποστολής Μινούς, ο κύριος Αμπτελαζίζ, θα μπορούσε να έλθει σε συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και να μας διαφωτίσει. Τέλος, επιμείναμε στον ρόλο τον οποίο η χώρα αυτή μπορεί να αναλάβει στη Μεσογειακή ε, Λεκάνη να θυμίσω ότι στις 25 Μαΐου ο δόκτωρ Ιουσέφ Μακράνη έγινε ο νέος Γενικός Γραμματέας της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Και αυτό προσθέτει θα έλεγα επιπλέον ευθύνες. Ξέρετε ότι το Μαρόκο αυτή τη στιγμή προεδρεύει στην εναλλασσόμενη Προεδρία της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης και προεδρεύει επίσης και του Ιδρύματος Αναλίντα Όλα αυτά είναι μεγάλες ευθύνες για την χώρα αυτή. Έχουν υπάρξει και πάρα πολλές αλλαγές βέβαια τον τελευταίο καιρό και θα πρέπει η προσπάθεια την οποία κάνει το Μαρόκο να μπορέσει να οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων που υπάρχουν. Και στα πλαίσια λοιπόν της Ευρωμεσογειακής και στα πλαίσια της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα της νέας πολιτικής γειτονίας και δεν θα πρέπει να αγνοηθεί το πρόβλημα από τα πολιτικά όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπουάιντα, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή των Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μας προσκάλεσε. Θα προσθέσω ακόμη δύο λόγια στα όπα, σε όσα δήλωσε ο κύριος Παντσέρη, λέγοντας ότι το κλίμα μας το οποίο διεξήχθησαν όλες τις συνεδριάσεις της Μικτής κοινοβουλευτική Επιτροπής ήταν καταρχάς κλίμα με μεγάλη ειλικρίνεια, το χαρακτηρίζει μεγάλη ειλικρίνεια και ανοιχτές τοποθετήσεις εκ μέρους των βουλευτών. Πιστεύω ότι φτάνουμε ως εκ τούτου σε ένα επίπεδο οριμότητας του διαλόγου υψηλό για τον διακοινοβουλευτικό διάλογο. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι κατά την συνεδρίαση για τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις, στην οποία ομάδα Μαροκινών αφενός και Ευρωπαίων αφετέρου βουλευτών ανέλαβε τη συντάξη εκθέσεως ε, έλαβε μέρος και το είπα το Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που είναι ανώτερη αναγνωρισμένη αρχή στο, Συμβου... στο Μαρόκο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι σήμερα την ώρα που εδώ σας παρουσιάζουμε την ε, έκθεση πεπραγμένων της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής το Μαρόκο ετοιμάζεται να ε, δεχθεί τον τίτλο «Ετέρος για τη Δημοκρατία» του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό αποτελεί για μας μεγάλη δέσμευση, διότι θα επιτρέψει την θεσμοθέτηση και την εδραίωση περαιτέρω του κράτους δικαίου με τους όρους και τα πρότυπα, τα διεθνή που θα θέλαμε να έχουμε και βέβαια να προχωρήσουμε προς ένα νέο σύνταγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Πρέντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη συνεδρία τη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου. Έλαβα και εγώ μέρος και θα ήθελα να σημειώσω τη ευχαριστία μου προς την κυρία Μποάιντα για την πολυθερμή υποδοχή. Το πρόγραμμα ήταν πολύ εντατικό. Ο κύριος Παντσέρος, πρόεδρος της προσωπία μας ε, για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέπ, περιέγραψε πολύ πιστά την ε, εξέλιξη των εργασιών. Θα ήθελα απλώ εγώ από πλευρά μου να επιμείνω σε δύο-τρία σημεία συγκεκριμένα που είχαμε στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων και που συζητήθηκαν με μεγάλη ειλικρίνη, όπως είπε και η συνάδελφος από το Μαρόκο. Είχαμε στην εμερή συνέταξη λοιπόν τη συζήτηση για την πολιτική μεταρρύθμιση, η οποία πιστεύω διεξήχθη κατά τρόπο πολύ ενδιαφέροντα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ο διάλογος μεταξύ των κομμάτων του Μαρόκου, κάθε πολιτικού χρώματος και βέβαια αντίστοιχα των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ο διάλογος ε, για την πολιτική μεταρρύθμιση, την πρόοδο στις δημοκρατικές, θέματα της δημοκρατίας. Ήταν ενδιαφέρουσα επίσης συζήτηση ως προς την ερμηνεία αλλά και την αμφισβήτηση που προκύπτει στο Μαρόκο. Και επίσης πολύ ενδιαφέρον ήταν, ε, πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η εξέλιξη στο Μαρόκο και σε άλλες χώρες του Μαγκρέπ μέσα σε μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων ειρηνική και όπου πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγης. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα και το οποίο ε, ανέλαβα εγώ με τον συναδελφό Απτελαχή Μαχμούν ε, το θέμα της περιφερειακής ολοκλήρωσης και το επισημαίνω γιατί είναι για το Μαρόκο θέμα μεγάλης σημασίας ευαίσθητο θέμα στην γενικότερη οικονομία της διαδικασίας των μεταρρυθμίσεων και γιατί βλέπουμε ξεκάθαρα τη βούληση να προσφερθεί, να προβληθεί μία λύση μαροκινή, μια λύση που να αφορά και να χαρακτηρίζει το Μαρόκο, βεβαίως πάντα σε αναφορά με τις διάφορες ε, προτάσεις και ιδέες διοικητικής οργάνωσης ευρωπαϊκές, αλλά ε, θέλουν βέβαια να βρουν τη λύση τη δική τους που θα σέβεται και θα ακολουθεί τις παραδόσεις ε, και την ιστορία του ήδη του Μαρόκου. Άρα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και επίσης τον έφερε ο κ. Παντσέρη, θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για την συνάντησή μας με τον κύριο Αμπτελαζή, Ανία Αμπτέλαζή, που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα επαφή. Μιλήσαμε δηλαδή με αυτό που αποκαλούν οι Μαροκινοί νότιες επαρχίες και είδαμε επιτόπου μαζί με τους υπεύθυνους αποστολή αυτής ε, το τι δραστηριότητες αναπτύσσονται τόπου. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος Παντσέρη, το κύριο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι η σταθερότητα και από την άλλη η ανάγκη για οργάνωση μιας απογραφής που θα επιτρέψει καλύτερη διαχείριση της κατάστασης. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα. Και ολοκληρώνω σημειώνοντας ότι οι ε, συναντήσεις με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, τους φίλους δηλαδή μαροκινούς συναδέλφους, αλλά και με εκπροσώπους κοινωνία των πολιτών, μας επιτρέπουν να σχηματίσουμε μια πολύ καλή εικόνα της επικαιρότητα στο Μαρόκο. Και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ποιότητα αυτού του διαλόγου, αυτής της ε, δουλειάς που έγινε στο πλαίσιο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μπεναραμπατσού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ήμουν μέλος αυτής της αντιπροσωπείας και είναι αλήθεια ότι είναι, ήταν ενδιαφέρουσες στιγμές. Έγιναν κάποιες ε, συζητήσεις έντονες, ε, τεταμένες, σε σχέση με την ε, θεώρηση διαβατηρίων και υπάρχει το έντονο αίτημα να επιτραπεί μια καλύτερη κυκλοφορία των ε, ανθρώπων να διευκολυνθεί δηλαδή η κινητικότητα. Ε, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το θέμα. Και κάτι άλλο. Σημαντική ήταν ε, η συνάντηση με τους ε, εκπροσώπους της ε, Il ε, ήταν σημαντικό και θεωρώ ότι πραγματικά είναι ενδιαφέρον ο ορίζον που διανοίγεται. Ε, είναι σημαντικό επίσης ε, το ζήτημα της αποκέντρωσης γιατί ε, με τον τρόπο αυτό μπορεί να λυθεί και το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας. Κάτι το οποίο με εξέπληξε είναι ότι υπάρχει ένα στίχος άμμου που οροθετεί την περιοχή και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές θαμένες νάρκες που προκαλούν πολύ συχνά ατυχήματα. Ε, πέφτουν θύματα χωρικοί αλλά και ζώα. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να οργανωθεί μια κοινή ομάδα με εκπροσώπους από τα δύο μέρη για να απομακρυνθούν αυτές οι νάρκες. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα βήμα προς την ενδεχόμενη συμφιλίωση. Δηλαδή να απομακρυνθούν οι νάρκες σε ολόκληρη αυτή τη ζώνη και από τις δύο πλευρές αυτού του τείχους της άμμου. Ε, το Μαρόκο επέτρεψε στους εταίρους μας του Νότου να συμβάλλουν στη διαδικασία εκδημοκρατισμού. Είναι μια ενδιαφέρουσα και σημαντική κίνηση που παρακολουθούν ενδιαφέρον και άλλες χώρες της Μεσογείου και του Μαγκρέμ. Πρόκειται για ένα ειρηνικό κίνημα, αλλά θα ήθελα να καλέσω τις αρχές να τείνουν ευήκο ους ε, προς όλες τις πλευρές στη ε, Ραμπάτ και σε άλλες ε, πόλεις ε, λαμβάνουν χώρα καθημερινά διαδηλώσεις, συνδικαλιστές, γιατροί κλπ. Το λαϊκό κίνημα της 20 Φεβρουαρίου είναι ιδιαίτερο ισχυρό και νομίζω ότι οι αρχές θα πρέπει πραγματικά να στρέψει την προσοχή τους προς αυτές τις κινητοποίησεις. Και υπάρχει ο κίνδυνος εάν δεν ληφθεί υπόψη το κίνημα αυτό από τις αρχές να υπάρξει στεναρή αντίσταση. Επίσης είναι αναγκαίο να λάβουν υπόψη οι εταίροι μας το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και της οικολογικής πολιτικής που μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος όλων των μέτρων τα οποία θα ελοπιθούν στην περιοχή όσον αφορά την οικονομία, τη γεωργία κλπ μιλήσαμε σχετικά με τους αρμόδιους υπουργούς και ε, θα ε, οι συνάδελφοί μας ε, από το Μαρόκο μας είπαν, μας είπαν στην προσοχή στο γεγονός ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην θέλουμε να τους δώσουμε μαθήματα. Είναι σημαντικό οι σχέσεις μεταξύ ερετών συναδέλφων στο πλαίσιο της πολιτικής της γειτονίας να αποτελέσουν ένα στοιχείο το οποίο να συμβάλλει στη διαμόρφωση διεθνών σχέσεων που να ανταποκρίνονται στο δικό μας ε, όραμα ως εκλεγμένων εκπροσώπων του λαού πέρα από τις πολιτικές των κυβερνήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπεναραμπάτο. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Παντσέρη να απαντήσει εφόσον το επιθυμεί. Σύντομα. Στο κλείσιμο λοιπόν της συζήτησης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη συμπροεδρό μου και τους ε, μαροκινούς εταίρους γενικότερα για την μεγάλη διαθεσιμότητα την οποία επέδειξαν και την υποδοχή τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας. Να ευχαριστήσω επίσης και τη Γραμματεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε μια συζήτηση χρήσιμη έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την τοπική πραγματικότητα στο ε, Μαρόκο και στην Ανατολική, στη Δυτική Μεσόγειο γενικότερα. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές δυνατότητες. Δεν πρέπει λοιπόν να μείνουμε στα λόγια. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την επιδίεξη των στόχων χωρίς να θέλουμε να είμαστε παρεμβατικοί, χωρίς να θέλουμε να μπλεχτούμε στα εσωτερικά άλλων χωρών. Το βασικό θέμα είναι ότι το να προλαμβάνει κανείς είναι προτιμότερο από το να θεραπεύει και θα πρέπει ακριβώς αυτές τις δημοκρατικές διαδικασίες να τις προωθήσουμε για να πετύχουν τους στόχους τους γενικότερα στις χώρες αυτές. Και σαν μεικτή επιτροπή διακοινοβουλευτική θέλουμε να συνοδεύουμε όπως μπορούμε χωρίς να θέλουμε να δώσουμε μαθήματα σε κανένα αλλά να βοηθήσουμε στο βαθμό του δυνατού. Καταλαβαίνω βέβαια αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Επιτροπή ΑΦΕΤ ιδιαίτερα για το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε το πλαίσιο λειτουργίας της αποστολής Μήνους για να υπάρξει μια γαλήνια συζήτηση γύρω από το θέμα. Όσο νωρίτερα γίνει αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις διαπραγματεύσεις που έχουν ε, ξεκινήσει στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι και η κυρία Μποάιντα. Απλά να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ λοιπόν όλους. Κλείνουμε με τη συζήτηση αυτή. Τώρα περιμένουμε την εξοχότητά του αντιπρόεδρο της Σερβικής Δημοκρατίας, τον κύριο Ντέλιτς. Θα είναι εδώ σε πέντε λεπτά. Διακόπτουμε λοιπόν για πέντε λεπτά. Παρακαλώ να επανέλθετε εγκαίρως. Λοιπόν, συνάδελφοι, έχουμε μαζί μας τον Αντιπρόεδρο κύριο Μπόζι Νταρντέλιτς, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κυβέρνησης. Είναι θα έλεγα συνηθισμένη η παρουσία του εδώ ευτυχώς και με μεγάλη χαρά για μια ακόμη φορά συναντώμεθα και θα συζητήσουμε ιδιαίτερα μετά από το τελευταίο σημαντικό συμβάν που μεσολάβησε, τη σύλληψη του Ράτκο Μλάντιτς, και την παρουσία του τώρα πλέον στη Χάγη, όπου θα δικαστεί για αυτά τα οποία κατηγορείται στη δεκαετία του 90 για τα οποία είναι υπεύθυνο λέω μιλητή στη δεκαετία του 90. Συναντηθήκαμε λοιπόν και με τον εκπρόσωπο της Προεδρίας λίγο πριν τον κύριο Μάτωνη. Ήταν ενθαρρυντική η συνάντηση αυτή, ιδιαίτερα στα θέματα της διεύρυνσης. Και είμαι βέβαιος ότι και εσείς θα μπορέσετε να μας δώσετε αρκετές λεπτομέρειες να τεθούν και ερωτήσεις από τους συναδέλφους και να διευκρινιστούν τα θέματα τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων. Έχετε το λόγο κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πάσκου. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, έχουν συμβεί αρκετά τους τελευταίους πέντε μήνες, από την τελευταία φορά δηλαδή που συναντηθήκαμε οι βασικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον Ράτκο Μλάντιτς. Αυτή ήταν η ηθική μας υποχρέωση και ήταν και ένα σημαντικό βήμα για την περιφερειακή συμφιλίωση. Δεν το κάναμε για να μας πει η Ευρώπη μπράβο ή για να μας ανοίξει τις πόρτες της. Πρέπει ακόμα να βρούμε τον Κόραν Χάτζιτς, θα συνεχίσουμε να καταπολεμούμε το οργανωμένο έγκλημα, θα συνεχίσουμε τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις μας. Ο στόχος μας για το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι ξεκάθαρος. Η άνοιξη του 2012 να οριστεί σαν στόχος στιγμής έναρξης των διαπραγματεύσεων. Η Κροατία ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις και το πέτυχε αυτό που είπαμε τώρα πριν 6 χρόνια. Δεν θέλουμε λοιπόν αυτό να είναι κάτι το χαριστικό, απλά εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς μας και το βασίζουμε στα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Όσοι είχαν πει τα τελευταία χρόνια ότι θα είναι σκληροί αλλά δίκαιοι με τη Σερβία, να τους πω συνεχίστε να είσαστε σκληροί αλλά μη γίνετε άδικοι. Μη γίνεται άδικη προς τους Σέρβους πολίτες εφόσον σεβόμεθα τα κριτήρια και μην εφευρίσκεται νέα εμπόδια τα οποία θα μπλοκάρουν το δρόμο για την Ευρώπη. Το να είναι κανείς αυστηρός είναι κάτι το καλό, αλλά το να είναι άδικος δεν είναι καλό. Και γι' αυτό λοιπόν αγαπητά μέλη, η συνάντηση αυτή είναι μια, ένα τμήμα θα έλεγα του ολοένα πιο εντατικού διαλόγου που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ο πρόεδρος Τάντιτς και ο πρωθυπουργός Μπέρκοβιτς συναντήθηκαν με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προηγούμενη εβδομάδα. Οι επαφές ε, είναι όλο και πιο συχνές λοιπόν και γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω στις 9 Σεπτεμβρίου να συναντηθούμε στα πλαίσια του πρώτου φόρουμ Ευρωπαϊκής Ένωσης Σερβίας το οποίο θα οργανώσουμε 300 εκπρόσωποι της πολιτικής ε, του επιχειρηματικού κόσμου ε, στον Δούναβη θα υπάρξει συνάντηση αυτή. Θα είναι παρόντες και οι πρόεδροι ε, κύριοι κύριοι Βαν Ρόμπαϊ και Τάντιτς. Ελπίζουμε να γίνει ένα ετήσιο λοιπόν ε, συμβάν αυτό το οποίο προγραμματίζουμε για το Σεπτέμβρη και ελπίζουμε εσείς να μπορέσετε να μας επισκεφτείτε γιατί η συνάντηση αυτή θα είναι χρήσιμη για όλους όσους παρακολουθούν την κατάσταση όχι μόνο στη Σερβία αλλά και στα Δυτικά Βαλκάνια. Αγαπητά μέλη λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη πλειοψηφία με την οποία στηρίξατε την εφαρμογή της συμφωνίας τον Ιανουάριο με τη Σερβία. 18 χώρες μέλη επικύρωσαν ήδη τη συμφωνία αυτή, αρκετές άλλες έχουν προχωρήσει, κάποιες όμως διστάζουν ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Το Μάρτιο έγινε μια, ένας μικρός ανασχηματισμός οι εκλογές, ε, οι βουλευτικές και οι δημοτικές θα γίνουν ταυτόχρονα την Άνοιξη. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά μας σε μια χρονιά και με εκλογές, προεκλογική περίοδο, αλλά και ε, συνέχιση της προσπάθειας μεταρρυθμίσεων. Μετά από το πράσινο φως τον προηγούμενο Οκτώβριο, ε, πράγματι σημειώθηκε ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Λάβαμε 2.500 ερωτήσεις και απαντήσαμε σε αυτές μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Πήραμε άλλες 639 ερωτήσεις το Μάρτιο και απαντήσαμε μέχρι τις 31 ε, Απριλίου. Υποδεχθήκαμε έξι αποστολές τεχνικές των κρατών μελών και της Επιτροπής και ήδη εφαρμόζουμε κάποιες από τις χρήσιμες συστάσεις τους. Εργαζόμαστε σκλήρα προσπαθώντας να αποδείξουμε αυτό που ονομάζεται στα έγγραφά σας διοικητική ικανότητα. Επί τη βάση του προγράμματος δράσης που υιοθετήσαμε τον προηγούμενο Δεκέμβριο, με στόχο την έναρξη των διαπραγματεύσεων είμαι πεπισμένος ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να παράσχουμε τη σωστή βάση ε, για να ε, μπορέσει να εκδώσει τη σύστασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασιζόμενη σε κριτήρια ουσίας. Όχι μόνο θα συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το να μας χορηγηθεί η ιδιότητα της υποψήφιας χώρας αλλά και θα προτείνει και ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων την επόμενη άνοιξη. Θέλουμε η γνωμοδότηση αυτή να ληφθεί, να αποφασιστεί με ομοφωνία. Να στραφώ τώρα σε έξι θέματα πάρα πολύ σημαντικά τα οποία ελπίζω να μπορέσουμε να πετύχουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Να μιλήσω για το ICPY, για την περιφερειακή συνεργασία, τις σχέσεις με την Πρίστινα, την, την δυνατότητα μετακίνησης χωρίς θεωρήσεις κτλ. Καταρχάς θα συνεχίσουμε την πλήρη συνεργασία μας με το Διεθνές Δικαστήριο για την Τέος Ιουκοσλαβία εμείς έχουμε παραδώσει ήδη 44 από τους 46 καταζητούμενους. Τώρα και ο Μλάντιτς μετά τον Κάρατζιτς ε, νομίζω ε, θα δικαστούν και αυτό αποδεικνύει την αξιοπιστία της κυβέρνησης Στάντιτς. Ο κύριος Μπούζεκ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, είπε ότι η σύλληψη του ε, Μλάντιτς είναι μια απτή απόδειξη της προσπάθειας και της βούλησης της Σερβίας και του σερβικού λαού. Και ο κύριος Βαν Ρόμπα είπε ότι ήταν κομβική η στιγμή αυτή και από εδώ και πέρα ανοίγει ο δρόμος. Μόνο η αλήθεια και η δικαιοσύνη και η αναγνώριση ευθύνης προσωπικής ή συλλογικής θα λύσει τα προβλήματα στην στα Βαλκάνια. Το ίδιο βέβαια θα πρέπει να συμβεί και για τα θύματα από πλευρά Σερβίας μετά από την έκθεση του Ντίκ Μαρτί για την παράνομη εμπορία ανθρώπινων οργάνων στο Πέδιο. Θα θέλαμε όλα αυτά τα θέματα να αντιμετωπιστούν μέσω των μηχανισμών που, προβλέπει, που προβλέπουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. εκδόθηκε, εκδόθηκε ένα ένταλμα σύλληψης για ένα Τούρκο πολίτη το οποίο όμως δεν έχει αυτή τη στιγμή εφαρμοστεί και ταυτόχρονα ο καταζητούμενος γιατρός λέει, δίνει συνεντεύξεις στον σερβικό τύπο λέγοντας ότι δεν κινδυνεύει να συλληφθεί. Το θέμα αυτό είναι σημαντικό για μας, γιατί ξέρετε ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης δεν ισχύει σε χώρες όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, το Μαρόκο κτλ. Απαιτείται ένας ad hoc μηχανισμός παράλληλα με το μηχανισμό του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εμείς δεν ζητάμε να συμβεί κάτι το διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που ήδη μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί. Δεύτερος τομέας είναι η περιφερειακή συνεργασία. Είναι βασική προτεραιότητα για μας. Το προηγούμενο Μάρτιο η Σερβική κυβέρνηση υιοθέτησε ένα ψήφισμα για τη Σρεμπρένιτσα. Ο πρόεδρος Τάντιτς ε, για δεύτερη φορά πήγε στη Σρεμπρένιτσα 15 χρόνια μετά από αυτή την τραγική σφαγή. Εμείς υποστηρίζουμε πλήρως την εδαφική ακεραιότητα της Βοσνίας Ευζεγοζίνης στα πλαίσια των συμφωνιών του Ντέιτον. Τον προηγούμενο Νοέμβριο ο πρόεδρος Ιωσίποβιτς και ο πρόεδρος Τάσδιτς πήγαν στο Βούκοβαρ και απότισαν φόρο τιμής και στους Σέρβους που έπασαν θύματα των πολεμικών, της διεξαγωγής του πολέμου εκεί. Το 2011 τυχαίνει και το 2012 η Σερβία ε, ήταν παρούσα σε πολλές ε, πρωτοβουλίες περιφερειακές, την κεντρικό, κεντροευρωπαϊκή πρωτοβουλία, την πρωτοβουλία της Αδριατικής και Ιωνίου και ε, στην, στην, στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας. Συμμετέχουμε στα προεδρία των οργανισμών αυτών, προσπαθώντας να λύσουμε τα περιφερειακά προβλήματα στα πλαίσια ενός νέου, ε, θα έλεγα παγκοσμιοποιημένου πλέον περιφερειακού συνόλου. Ε, κάποια πράγματα έχουν πάει καλά, πολλά λουλούδια έχουν ανθίσει, υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες όμως και η Σερβία μόνη της δεν μπορεί να τις λύσει στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας να αναφερθώ σε μια πρωτοβουλία σερβική με άλλες χώρες χωρίς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα έγγραφο που σας μοιράζουμε σήμερα και παρουσιάζει την κοινή θέση για τις δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2013. Βλέπουμε ότι τα προγράμματα αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δίνουν πάνω από το 1% για την διεύρυνση στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Σήμερα είναι 1,3 με 1,4. Γνωρίζοντας ότι κάποιες από τις ιδέες τις οποίες έχει υιοθετήσει το κοινοβούλιο σας το σύνολο του κοινοτικού προϋπολογισμού φέρεται ότι δεν θα πρέπει να είναι πάνω από το 1% του συνολικού ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα της διεύρυνσης που έχει τόσο συζητηθεί δεν θα πάρει πάνω από 0,01% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δείχνει το επίπεδο προτεραιότητας το οποίο αποδίδεται στην διεύρυνση. Όχι, δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επαναξιολογήσουν τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Γνωρίζοντας το τι έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν και γνωρίζοντας τα αμοιβαία πλεονεκτήματα όπως α, στρατηγική του Δούναβη ας πούμε τον διάδρομο υπαριθμών 10, οδικό και σιδηροδρομικό, ωφέλιμο για όλους. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε τρένα τα οποία να πηγαίνουν με 120 χιλιόμετρα γιατί αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάει κανείς από την Βιέννη ή τη Βουδαπέστη στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά από την άλλη από μόνοι μας δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς των 120 χιλιόμετρων την ώρα αν δεν αλλάξει κάτι στα πλαίσια αυτών των δημοσιονομικών προοπτικών. Είμαστε λοιπόν ρεαλιστές και αυτό το οποίο προτείνουμε σε αυτή τη φάση στα πλαίσια των μηχανισμών των δημοσιονομικών προοπτικών να αναγνωρίσετε κάποια από τα προβλήματα που έχουν μείνει από το παρελθόν για τις χώρες στην διαδικασία ε, ε, διεύρυνσης ε, οι πόροι που είναι διαθέσιμοι τώρα είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Για τη Σερβία 190 εκατομμύρια κατέτος και το 70% ποτέ δεν φτάνει στη Σερβία γιατί πληρώνεται σαν περντίεμ σε συμβούλους οι οποίοι μας επισκέπτονται. Εάν λοιπόν θέλουμε να βάλουμε μια ευρωπαϊκή σημαία για κάπτη στην Σερβία, για μια μικρή γέφυρα, για ένα συλλέκτη νερού, για ένα σχολείο, για, ε, για έναν συνοικισμό Ρωμά, τότε χρειαζόμαστε 30 με 40 εκατομμύρια τον χρόνο. Ας πάρουμε το παράδειγμα της Κροατίας. Πέρνα, θα περάσει από 150 εκατομμύρια μέσα σε λίγους μήνες σε δύο δις κατ' Λοιπόν, λίγα στην αρχή για να προετοιμαστεί, πάρα πολλά μετά για να απορροφηθούν. Λοιπόν, δεν λέμε ότι οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες της ε, ένταξης από τη μία της διεύρυνσης και τις χώρες μέλη από την άλλη θα πρέπει να, ε, να μην υπάρχουν. Είναι προφανές ότι θα υπάρχουν, αλλά διαφορές 1 προς 10 ή 1 προς 15 θεωρούμε ότι δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος και θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα τα επόμενα χρόνια γιατί θα υπάρξουν ε, μετά την ένταξη της Κροατίας δεν θα υπάρξουν εύκολα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Δυτικά Βαλκάνια μετά το 2013 θα απομονωθούν και πολιτικά και οικονομικά και δημοσιονομικά. Εμείς δεν ζητάμε πάρα πολλές μεγάλες αυξήσεις, αλλά μια γραμμική αύξηση της στήριξης και εφαρμογή της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να υπάρξει μια επιλεκτική κατανομή των πιστώσεων αυτών. Εμείς ε, δεν μας λείπουν πράγματα τα οποία μπορούμε να εξηγήσουμε ότι είναι χρήσιμο να προωθηθούν. Τα Δυτικά Βαλκάνια δεν ζητούν ούτε ένα ευρώ ε, ε, για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν αυξήσαμε τους φόρους, μειώσαμε τις δαπάνες, και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα που δεν ξεπερνάει το 4% του ΑΕΠ. Το εξωτερικό μας χρέος είναι 43% πολύ πιο κάτω από τα κριτήρια του Μάστρι. Αν δει κανείς όμως τις προοπτικές μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα δει ότι δεν υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης αν δεν αλλάξει τίποτα στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν τα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά και τότε δεν θα υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχουμε ε, σε ε, έργα υποδομών ευρωπαϊκά σαν παράδειγμα να χρησιμο... πείτε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την, τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα τα καταφέρουμε γιατί δεν εντασσόμεθα στα κριτήρια τα οποία απαιτούνται και δεν μπορούμε να πάρουμε μέρος σε μελλοντικές ευρωπαϊκές προσπάθειες όπως οι υποδομές, τις μεταφορές ή η προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα κτλ. Εάν τα ποσά τα οποία χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να αυξηθούν, ίσως θα υπάρξουν περισσότερα προβλήματα στον τομέα της γεωργίας και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάποιες επιλογές. Μια δεύτερη ιδέα που θα βρείτε στο έγγραφο αυτό και είχα την δυνατότητα να τα παρουσιάσω αυτά στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι τα Δυτικά Βαλκάνια να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αντιπροσωπεύει στους προϋπολογισμούς τα ποσοστά και μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τις ευρωπαϊκές εγγυήσεις στις δυνατότητες πρόσβασης που έχει στις διεθνείς χρωματαγορές. Ε, τα Δυτικά Βαλκάνια ε, θα πετύχουν πολλά αν στηριχθούν με αυτόν τον τρόπο και σε επίπεδο μακροοικονομικό και θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει σαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να μας βοηθήσει να έλθουμε σε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ηλικίε συνταξιοδότησης οι οποίες να είναι υποστηρίξιμες και με γενικότερα επίπεδα αμοιβών τα οποία να μην είναι λαϊκιστικά. Είναι δηλαδή ε, πολιτικές οι οποίες θα μας ωφελήσουν εμάς αλλά θα ωφελήσουν συνολικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς λοιπόν θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σας και στον τομέα αυτό. Τρίτον, θέλουμε να πιέσουμε για έναν πιο κακοφόρο διάλογο με την Πρίστινα. Εμείς έχουμε προτείνει ένα διάλογο με την Πρίστινα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, προτείνοντας ε, ένα κοινό ψήφισμα το οποίο έγινε δεκτό διαβοής. Έχουν ήδη υπάρξει τέσσερι γύροι διαπραγματεύσεων, έχει υπάρξει πρόοδος και στα θέματα των μητρών και στα θέματα του κτηματολογίου, της ελεύθερης διακίνησης και των δικτύων ηλεκτρισμού. Θέλουμε να υπάρξει περαιτέρω πρόοδο σε σχέση με τα τέλη, τα τελωνιακά, Μικρά βέβαια βήματα προόδου, αλλά παρόλα αυτά μετά από τόσα χρόνια εντάσεων και βίας είναι θετικά. Ο διάλογος με την Πρίστινα θα οδηγήσει, ελπίσουμε, σε κάποια φάση στον ιστορικό συμβιβασμό ανάμεσα στους ε, κατοίκους του Κοσφοπεδίου και τους Σέρβους. Οποιαδήποτε άλλη λύση δεν είναι δυνατή και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσφοπεδίου. Θέλουμε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να βρούμε μια κάποια λύση πριν γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πρίστινα χρειάζεται αυτή τη συμβιβαστική λύση ακόμα περισσότερο και αυτό είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σχέση λοιπόν με το συγκεκριμένο θέμα εμείς δεν, δεν υπαναχωρούμε, δεν κάνουμε αντίσταση θα έλεγα, έχουμε στραφεί προς τα εμπρός και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να βρεθεί λύση σε όλα τα θέματα, ακόμα και στα πιο δύσκολα, τα οποία θα ανοίξουν ένα ευρωπαϊκό μέλλον σε όλους τους πολίτες. Τέταρτον, εμείς θέλουμε να διατηρηθεί το ε, καθεστώς ε, της ε, κυκλοφορίας με ελεύθερες θεωρήσεις. Άνω των 6 εκατομμυρίων ε, περασμάτων σε εισαγωγικά Σέγγεν έχουν συμβεί από τότε που θεσπίστηκε το καθεστώς αυτό. Πάνω από 3 εκατομμύρια Σέρβων έχουν βιοματρικά διαβατήρια, έχουν υπάρξει 6 λοιπόν ε, εκατομμύρια περάσματα και υπάρχουν 17.000 Σέρβοι οι οποίοι έχουν καταγραφεί ως ετούντες πολιτικό άσυλο στην Γερμανία, στην Αγγλία. Άνω του 90% των ετοιμάτων έχει απορριφθεί. Έχει υπάρξει 40% μείωση σε αυτούς οι οποίοι ζητούν άσυλο σε όλες τις χώρες ανάμεσα στον προτελευταίο και τον τελευταίο χρόνο. Δημιουργήσαμε μια διυπουργική επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρμογής του καθεστώντος Σέγγεν έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα αυτούς οι οποίοι ε, οργανώνουν ε, αυτούς οι οποίοι ζητούν άσυλο, οργανώνουν ομάδες τον άσυλο και θα συνεχίσουμε εμείς τον ε, αυστηρό έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων, θα το κάνουμε αυτό χωρίς σε καμία περίπτωση να δακτυλοδεικτούμε η αδίποτε φιλετική ομάδα σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στις ευέλωτες ομάδες ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα και δεν θα επηρεαστούν οι διαδικασίες για την χορήγηση πολιτικού ασύλου όπου αυτό χρειάζεται και αυτό ισχύει και για τους Ρωμά και άλλες κοινότητες. Θεωρούμε ότι είναι θετικές οι προτινόμενες αλλαγές στους κανόνες του Σέγγεν, και οι κυρώσεις που επιβάλλονται με την απαγόρευση σαν παράδειγμα ε, ε, εκ νέου συνόδου στην περιοχή ε, Σέγγεν για κάποια χρονικά διαστήματα. Στην Νορβηγία έχουμε ένα παράδειγμα, ο αριθμός αυτών οι οποίοι αιτούνται ασύλου ακριβώς ο αριθμός τους από 20.000 σε κάποια φάση έχει μειωθεί τώρα σε ε, ένα ελάχιστο αριθμό, 19 μόνο αν ακούσαμε καλά. Εν πάση περιπτώσει αυτό έγινε με το νέο τρόπο επεξεργασίας της αίτηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτρέπει αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πραγματική ανάγκη. Όλα αυτά λοιπόν έχουμε προσπαθήσει έχουμε συνεργαστεί και τα έχουμε πετύχει. Έχουμε πολλαπλασιάσει τις επιχειρηματικές επαφές. Πολλές γιαγιάδες πηγαίνουν να βοηθήσουν τα εγγόνια τους όταν αρρωσταίνουν από τη Σερβία στη Γερμανία όταν αυτό χρειάζεται και όλοι έχουμε μια εικόνα της Ευρώπης η οποία δεν ελέγχεται από τους πολιτικούς και τα μέσα ενημέρωσης αλλά έχουν μια άμεση εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση που δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι απαιτούν να εργαστούμε σκληρά αλλά αποδεικνύει επίσης η εικόνα αυτή ότι και κανείς δεν είναι εναντίον μας χωρίς λόγο και άδικα. Λοιπόν, αυτό αυτές οι ελεύθερες μετακινήσεις χωρίς θεωρήσεις είναι ένα μεγάλο δώρο και θα συνεχίσουμε να το χαιρόμαστε. Η κυβέρνησή μας παράλληλα έχει υιοθετήσει και ένα πρόγραμμα δράσης για τις μεταρρυθμίσεις. Τώρα δεν θα αναφερθώ στα 96 σημεία αυτού του προγράμματος δράσης. Αλλά μετά από μια πρώτη τρίμηνη θα έλεγα αξιολόγηση Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μια συνάντηση στα πλαίσια του προωθημένου διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κάνουμε και την πλήρη αξιολόγηση μέσα σε λίγες εβδομάδες. Θα σταθώ όμως σε τέσσερα θέματα. Μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό, καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, μεταρρύθμιση επίσης ε, του ε, συστήματος της δημόσιας διοίκησης. Καταρχάς για το δικαστικό σώμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Το είδαμε στις χώρες οι οποίες γίνονται νέα μέλη ότι το θέμα αυτό είναι το σκληρότερο να αντιμετωπιστεί. Υιοθετήσαμε το Δεκέμβριο μία σειρά νόμους ε, επί τη βάση των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας. Τα μόνιμα μέλη του υψηλού του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου αποτελούνται πλέον κατά 97% από δικαστές και εισαγγελείς. Συμφώνησαν τον προηγούμενο μήνα στις διαδικασίες μέσω των οποίων θα αναθεωρήσουν κάθε απόφαση για διορισμό δικαστών και αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο φθινόπωρο. Συνεδριάζει η Επιτροπή αυτή μερικές φορές για 13 ώρες για να μπορέσει να καταλήξει σε αποφάσεις οι οποίες να είναι αποδεκτής για όλους γιατί ασκήθηκε δικαιολογημένη κριτική και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ίδιους τους δικαστές. Για τη διαφθορά δεν θα αναφερθώ στον αριθμό των ανθρώπων που συνελήφθησαν, δεν είναι ευχάριστο αυτό. Προχωράμε όμως για το οργανωμένο έγκλημα. Ήδη τον προηγούμενο μήνα στην Βραζιλία η μυστική αστυνομία μας σε συνεργασία με τις αστυνομίες των κρατών μελών και της Βραζιλίας έσπασε ένα μεγάλο καρτέλ ναρκωτικών. Στο θέμα το εκλογικό ε, τα ομαδικά ψηφοδέλτια ε, έχουν ε, επιληθεί σαν πρόβλημα και το Κοινοβούλιο δέχτηκε και μία τροπολογία έτσι ώστε από του χρόνου να υπάρχει τουλάχιστον κατά το 1 τρίτο παρουσία γυναικεία στο Κοινοβούλιο. Και έτσι φτάνουμε πάνω από τα απαιτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν και για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα είχα μία συνάντηση με οικογένειες παλαιών ιδιοκτητών. Συναισθάνεται κανείς την αδικία που είχαν ζήσει στην περίοδο του 1958 θα υπάρξει μία λύση ήδη μέχρι τον Σεπτέμβριο, μία πρώτη πρόταση τον Ιούλιο και η πρόταση αυτή θα γίνει αντικείμενο συζήτησης με τους άμεσα ενδιαφερομένους, αυτούς που είχαν χάσει τα σπίτια τους, αλλά φυσικά θα έρθουμε σε επαφή και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, όταν μιλάμε για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, είπα ότι τα ελλείμματά μας και το χρέος μας είναι χαμηλά. Η επένδυση της Fiat ενός δις για την παραγωγή 250.000 το 2012 έχει προχωρήσει Επίσης και η εταιρεία Deleuze θα αγοράσει το σύνολο των μετοχών του λιανεμπορίου μας. Έχουμε επίσης ε, γερμανικές εταιρείες που επενδύουν στη χώρα μας, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, Κορεάτες, Σλοβαίνους και νομίζω ότι έχουμε συνολικά έναν στόχο για τον χρόνο αυτό γύρω στο 3 με 4 δις. Έχουμε όμως κοινωνικό κόστος. 19,26% η ανεργία. Και εδώ υπάρχουν τρομερές διαφορές ανάμεσα στις περιφέρειες και ανάμεσα στις γενναίες. Η φτώχεια ε, ε, ανάμεσα στο 2003 και το 2008 είχε πέσει αλλά τώρα ξανανέβηκε όμως τα τελευταία χρόνια και υπάρχει πολλοί κόσμος που, ζουν, ε, που ζει με 2.000 ευρώ την ημέρα με 2, με 2 ευρώ συγγνώμη την ημέρα Έχουμε πάρα πολλά λοιπόν να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να μεταρρυθμίζουμε τα συστήματά μας, θα συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις υποδομές, θα κατασκευάσουμε τρεις γέφυρες στο Δούναβι και μία γέφυρα στον ποταμό Σάβα, ολοκληρώνουμε τον αυτοκινητόδρομο του διαδρόμου 10 και έχουμε κάνει και σημαντικά βήματα στον τομέα της ενέργειας ε, είχαμε συνάψει συμφωνίες την προηγούμενη εβδομάδα με Καναδούς και με την ΕΝΙΤ της Ιταλίας για τα υδροηλεκτρικά μας ε, εργοστάσια. Συμπερισματικά το 2011 θα είναι μια καταληκτική χρονιά για τις προσπάθειες της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων. Η Σερβία παρά τις δυσκολίες κινείται. Θέλουμε να αξιολογηθούμε όπως όλες οι άλλες χώρες επί τη βάση των θετικών μας επιδόσεων. Εμείς εφόσον μας δώσετε τη δυνατότητα θα λειτουργήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αν μας δώσετε μία ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό θα είναι πραγματικά σαν να έχουμε κερδίσει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι μπορούμε να υπολογίζουμε στη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είστε αυστηροί αλλά να είστε δίκαιοι. Για μια ακόμη φορά λοιπόν είμαι πολύ ευχαριστημένος που σας συνάντησα και ελπίζω να συναντηθούμε πάλι το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι για να δούμε τις δυσκολίες που μένουν αλλά και τις προσπάθειες που έγιναν. Well, Deputy Prime Minister. Κύριε Αναπληρωτή Πρωθυπουργέ, σε συγγνώμη γιατί αντί για Τζέλιτς είπα Και ξέρετε, εμεί στη Ρουμανία όταν κάνουμε τέτοιο λάθος, ε, λέμε ότι χρωστάω αρνή, χρωστάμε αρνή στον άλλον. Γι' αυτό λοιπόν σας χρωστάω ένα αρνή. Επισημάνατε θέματα οικία σε μένα, ιδίως το μοτίβο αυστηρότητα αλλά δικαιοσύνη μου είναι πολύ οικείο. Θα δούμε τι θα γίνει και μετά τι συνεδρίαση και σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Να δούμε. Ελπίζουμε ότι αν φτάσουμε μέχρι εκεί θα βρεθεί και κάποιος να μας υποδεχθεί. Ο κύριος Κούκαν τώρα, επικεφαλής αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρακαλώ να λάβει το λόγο για τρία λεπτά. Είναι ο μόνος ο οποίος θα έχει τρία λεπτά χρονομιλίας, οι άλλοι συνάδελφοι δύο λεπτά μόνο. Ξέρετε ότι έτσι γίνεται όταν δεν έχουμε χρόνο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ αναπληρωτή Πρωθυπουργέ, κύριε Πρεσβευτά. Θα ήθελα να επισημάνω ότι με το ψήφισμα των ΗΕ για την κατάσταση του Κοσφοπέδιου μπορέσατε να κερδίσετε σημαντικό και ούριο άνεμο στα πανιά του ευρωπαϊκού σας πλοίου και είσαστε στη σωστή κατεύθυνση. Η παράδοση του Μλάντετς στο δικαστήριο της Χάγης αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Μία παρατήρηση μόνο, καταγράφοντας τις αντιδράσεις των πολιτικών από πλευράς Βελιγραδίου, για ένα δευτερόλεπτο, μόνο για ένα δευτερόλεπτο όμως, μου δόθηκε η εντύπωση ότι ε, υπερέβαλαν τη σημασία αυτού του βήματος. Μετά όμως ε, ε εγκατέλειψα την ιδέα αυτή γιατί θα ήταν λάθος το συμπέρασμα. Ήταν αντίθετο πολύ σημαντικό το βήμα και ανοίγει το δρόμο για πιο γρήγορη πρόοδο, αλλά ασφαλώ όχι για τα πάντα. Θα πρέπει να ετοιμαστείτε για την μακρά, δύσκολη και περίπλοκη περία, πορεία προ τι ευρωπαϊκέ διαπραγματεύσει. Να πάρει το καθεστώ ψήφιου κράτου, ημερομηνία για την άνοιξη των διαπραγματεύσεων, των διαπραγματεύσεων. Είναι θέματα δύσκολα, δηλαδή θα πρέπει να προξενείτε φρούδες ελπίδες στον λαό σας ότι τα αυτά θα συμβούν πολύ γρήγορα και θα πρέπει να είσαστε προετοιμασμένοι ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολα από ό,τι μπορεί να περιμένετε όλα αυτά. Και όπως έλεγε και ένας Αμερικανός στρατηγός, μέχρι να τελειώσει δεν έχει λήξει. Και σας ε, προτείνω λοιπόν, ξέρετε τι έχετε να κάνετε, έχετε τα οράματα, έχετε τα σχέδια, τα χρονοδιαγράμματα στη διάθεσή σας, τα πάντα. Όπως ξέρετε, εμείς πάντα προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Είστε πια στο δρόμο της επιτυχίας. Δεν θα πρέπει να μειώσετε τις επιδόσεις, αντιθέτως να τις ενισχύσετε. Και σε όλα τα θέματα που αναφέρατε, διάλογο με το κοσφοπέδιο, περιφερειακή συνεργασία και το καθεξής, δεν μπορώ να σας πω, έχετε μπει στο σωστό δρόμο. Και ελπίζω να προχωρήσετε με επιτυχία όπως από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Κουκάν. Κυρία Μπράθνερ, παρακαλώ. Για δύο λεπτά. Uh, Πρόεδρε, δεν ακολουθούμε τη σειρά των συντονιστών. Είναι σκιώδες. Α, όχι, γιατί νόμιζα ότι εμεί προηγούμαστε των πρασίνων. Όχι, όταν μιλούν οι σκιώδει δεν έχουμε θέματα προτεραιότητα. Κύριε Μπράτνα. Σημειώνουμε, γνωρίζουμε ότι είμαστε η πέμπτη σε μέγεθο ομάδα, μην ανησυχείτε. Χαίρετε κύριε Τίλιτς, καλώς ήρθατε, με χαρά σας ξαναβλέπω και Συγχαρητήρια και για την σύλληψη και την παράδοση του Μλάντιτς. Ήμασταν πάντα πολύ αυστηροί στο θέμα αυτό και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε ότι ήμασταν και δίκαιοι γιατί σας συγχαίρουμε τώρα για αυτό το μεγάλο βήμα όπως το βλέπουμε εμείς το οποίο σας φέρνει πολύ μπροστά σας, δίνει μεγάλη όθηση. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τα λόγια σας ε, για τη δουλειά αυτή που γίνεται βέβαια και ο οργανισμός ε, για την προστασία των γυναικών να κάνει από πλευρά του μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. φυσικά θα πρέπει να βρείτε την χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό σας, αλλά πάντως έχει μεγάλη σημασία και έχετε πολύ καλές επιδόσεις. Σε σχέση όμως με το λαθρεμπόριο οργάνων για μεταμόσχευση. Είπατε ότι θα πήγαινε στα Ηνωμένα Έθνη. Μα πήγε ήδη στα Ηνωμένα Έθνη και το έκλεισε η Κάρλα Τελπόντε. Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλετε να επανέλθει το θέμα αυτό στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν έχει ίσω και τόσο μεγάλη σημασία για τη διεθνή ασφάλεια. Και ναι, μεν δεν αναγνωρίζετε την Όιλεξ, αλλά μήπως ήταν σκόπιμο να υποστηρίξετε το έργο της, γιατί δεν βλέπω σε τι θα σα βοηθούσε να ξαναστραφείτε προς τα Ηνωμένα Έθνη. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μερικές φορές ακολουθεί τη σειρά των συντονιστών, μερικές φορές μια τυχαία σειρά. Εν περιπτώσει, ξέρετε ότι είμαστε υπερήφανοι τώρα που είμαστε πιο πολύ από τους πράσινους, μην το ξεχνάτε. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ τον κύριο Ντέλιτ, να τον συγχαρώ εκ μέρου τη ομάδα των στρατικών δημοκρατών, και ιδιαίτερα για τη σύλληψη του στρατηγού Μλάντιτ. Αυτό αποτελεί πιστεύω ένα μεγάλο βήμα στο δρόμο του κλεισίματος ενός ζωφερού κεφαλαίου και θλιβερού στην ιστορία του λαού σας. Πιστεύω ότι μπορείτε να προχωρήσετε πολύ γρήγορα, έχετε κάνει μεγάλο μέρος της δουλειάς και για τις προοπτικές ως μόνιμος ε, εισηγητής για το Μαυροβούνιο που αισθάνεται μεγάλη απογοήτευση και αίσθημα ματέωσης διότι δεν έχουν λάβει ακόμη καμία ένδειξη για έναρξη διαπραγματεύσεων θα έλεγα ότι θα ήταν καλό η Επιτροπή να προσαρμόσει στην ίδια ευθεία να ευθυγραμμίσει το Μαυροβούνιο τη Σερβία και την Μακεδονία έτσι ταυτόχρονα να τους δώσει ε, ημερομηνία για έναρξη διαπραγματεύσεων κάπως αρχές του προσεχούς έτους ε, εάν βέβαια είναι δυνατόν αυτό. Φυσικά και θεωρώ ότι θα πρέπει κάθε χώρα να εξετάζεται εάν είναι καλή να ξεκινήσει διαπραγματεύσει τη ε, την ίδια ε, αυτόνομα, ε, αλλά παρόλα αυτά ίσω θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει αυτή η ευθυγράμμιση. Βέβαια, πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ενοχλημένο ότι όσο ότι η Μακεδονία και τι έχει κάνει τόσο μεγάλη πρόοδο, δεν επιτρέπεται να ανοίξει διαπραγματεύσει λόγω των διμερών σχέσεων με γειτονικό τη κράτο. Εν πάση περιπτώσει ελπίζουμε ότι η Κροατία, το προσεχές από ό,τι φαίνεται, κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα βοηθήσει και αυτή από πλευρά της. Σε ποιο βαθμό λοιπόν ε, μπορεί να ενισχύσει ή και να ε, καθυστερήσει, να δημιουργήσει δυσκολίες στην πορεία σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κροατία και βέβαια για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και κάτι άλλο, μια και εγώ θεωρώ το κοσφοπέδιο είναι σκόπιμο εδώ και καιρό μάλιστα υποστηρίζω την ιδέα τη απόσχηση του κοσμοπεδίου και με μεροληπτικό στο ξέρω, αλλά αυτά θα ρωτήσω το Υπουργείο των Εσωτερικών σα τι κάνει και σε ποιο βαθμό επιτρέπει την εκπροσώπησή του στου διεθνεί οργανισμού. Γιατί μέχρι να γίνει αυτό δεν μπορεί να υπάρξει μια οριστική ρύθμιση του ζητήματο του κοσμοπεδίου. Πρέπει να βρεθούν λύσει δημιουργικέ και εφάνταστε για να τελειώσει, για να λήξει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, κύριο Βάγκελ. Δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Ντέλιτς, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που ήρθατε να συζητήσουμε τις ευρωπαϊκές προοπτικές της Τουρκίας, της ε, Σερβίας, συγγνώμη, σε μια χρονική στιγμή όπου έχετε πια απαλλαγή από το μεγάλο αγκονάρι που κουβαλάγατε. Όλοι ξέρουμε ποιο ήταν, δεν μπορούμε να το επιβεβάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ε, θα ήθελα να ενισχύσω τις προσπάθειές σας και την δική σας μη άλλο επιλογή να μιλάτε πάντα για την μοντέρνα Σερβία, όχι τα, τα προ-μοντέρνα ή μετα-μοντέρνα αλλά τη μοντέρνα Σερβία. Και θυμάμαι την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει, ε, είχαμε πει ότι θα πρέπει ο σερβικός λαός ε, να αντιληφθεί ότι ο Μλάντιτς δεν ε, περιποιεί τιμή, αλλά ντροπή στη Σερβία, όνειδος και ήρθε πλέον η στιγμή η Σερβία να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κράτος. Πολλά μένουν να γίνουν. Έχετε ήδη χαράξει το δρόμο με το κυβερνητικό σας πρόγραμμα και τους προσανατολισμούς, νέες επενδύσεις, άνοιγμα προς το εξωτερικό. Εμείς βοηθούμε από πλευράς μας με το καθεστώς ε, αποδέσμευση από την υποχρέωση ε, θεώρηση διαβατήριων. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως, γιατί μιλάτε για κοσμοπέδιο μόνο, όχι για Πρίστινα, δεν θα έπρεπε να είναι αυτό το επόμενο βήμα. Εμείς αυτό περιμένουμε να δούμε. Και πρέπει ο πολιτικός λόγος που εκφράζεται να είναι ρεαλιστικός, γιατί αυτό θα απέβαινε εις όφελός σας, καθώς επίσης πιστεύω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό η Σερβία να εξακολουθήσει να διαδραματίζει επικοδομητικό ρόλο στην περιφέρειά της, Δηλαδή τόσο στο Μαυροβούνιο όσο και στη Βοσνία Αρσεγοβίνη, εκεί δηλαδή όπου ζουν Σέρβοι, εκεί όπου το Βελιγράδι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό πολιτικό ρόλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σερ Ρόμπερτ. Ευχαριστώ. Α είμαι ειλικρινή, αν μου επιτρέπετε, και να ζητήσω ταχύε απαντήσει, γιατί να σα εμπιστευτούμε όσον αφορά την κατάσταση των εγκληματιών πολέμου δεδομένου ότι πληρώνεται τη σύνταξη του Μπλάντιτς για τόσο καιρό. Δεύτερον, φαίνεται ότι η σερβική κοινή γνώμη αρνείται τις φρικαλαιότητες και υποστηρίζει τον Μιλόσεβιτς και επίσης υποστηρίζει τον Μπλάντουτς σε σχέση με αυτό το οποίο έπραξαν. Τρίτον, ακολουθώντας αυτά που είπε ο νεότερος συνάδελφός μου προηγουμένως, θα ήθελα να πω το εξή. Πώς ε, θα βοηθήσει αυτό τις σα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν γίνετε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς θα μπορέσετε να αντιδράσετε προς την Κροατία γιατί είδαμε κάποια προβλήματα στο τρόπο που η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπροι ανησυχούν ε, σε σχέση με την ε, Τουρκία και κάνουν την ε, ζωή δύσκολη στην Τουρκία όσον αφορά την αίτηση προσχώρησης. Τέλος, το ζήτημα του Κωσυφοποδίου. Είπατε ότι θα πρέπει να επιληθεί. Πώς όμως, αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Είναι ένα κομμάτι βρετανικής αισιοδοξία αυτό το οποίο εκφράσατε. Τώρα ο κύριος Νικολάη, η κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, εκ μέρους του Άλντε θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ και θα ήθελα να σας ε, εξασφαλίσω, να σας διασφαλίσω ότι η ομάδα μας υποστηρίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας σας και των Δυτικών Βαλκανίων. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη θα ολοκληρωθεί με σας και το εγχείρημα αυτό θα σευθεί με επιτυχία εφόσον προσχωρήσετε και εσείς στην Ευρώπη. Έχω μία ερώτηση η οποία σχετίζεται με το πρόγραμμά σας και θα ήθελα να σας ομολογήσω ότι υπάρχουν πολλοί εδώ που θεωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις που κάνετε στη Σερβία δεν είναι πραγματικά αρκετά σοβαρές. Εγώ ειλικρινά πιστεύω στη σοβαρότητα των μεταρρυθμίσεών σας γιατί βλέπω τα αποτελέσματά τους και μπορώ να τις συγκρίνω με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει σε άλλες χώρες μέλη. Και εσείς ε, πιστεύω είστε ένα πετυχημένο παράδειγμα αυτού του είδους των μεταρρυθμίσεων. Τώρα μια άλλη ερώτηση σχετίζεται με την αντίδραση της κοινή γνώμης στη σύλληψη του Μπλάντιτς. Πείτε μου, πόσο ε, σοβαρές είναι αυτές οι αντιδράσεις των ε, Σέρβων πολιτών. Και θα ήθελα να σας πω ότι υποστηρίζουμε πλήρως ε, τα όσα είπατε σε σχέση με τον προπολογισμό. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δείξει ότι η εξωτερική πολιτική θα είναι μια μείζον πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να διατηρήσουμε τα ποσοστά τα οποία δίδονται για αυτό το ζήτημα. 1,3 ή 1,5 μπορούν να εξασφαλίσουν αυτή την πολιτική και να καταδείξουν αυτή την πολιτική βούληση. Το άλλο ερώτημα σχετίζεται με τη στρατηγική του Δούναβη. Ποιο είναι το δικό σας όραμα εδώ. Ο κύριος Χόιτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ Ελπίζω ε, να χαρείτε τις ε, συζητήσεις ε, εδώ στο Κοινοβούλιο Σας εύχομαι καλή επιτυχία για τον πρωταθλητή σας στο τένις. Τώρα, όσον αφορά τι προοπτικέ για τη χώρα σα θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω τα όσα είπατε σήμερα το πρωί, σαν μια χώρα η οποία ήταν πολύ σκληρή στη σύλληψη των εγκληματιών πολέμου. Ε, κρεμεί η σύλληψη του χάτζη. και βεβαίως θα πρέπει να λάβουν χώρα διώξει όλη την περιοχή. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η σύλληψη των Πλάντιτς υπό την έννοια αυτή, να λειτουργήσει πραγματικά και ε, πραγματικά σας συγχαίρω. Τώρα, όσον αφορά το κοσυφοπαίδιο, είπατε ε, θα υπάρξει εδώ μια ελπίζω ότι θα ε, μπορέσετε να πετύχετε μια πρόοδο και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Τώρα, σε κάθε χώρα της περιοχής υπάρχει ένα πρόβλημα της Ρωμά. Στη δική σας, δική σας χώρα παλεύουμε το θέμα αυτό όπως και όλες οι άλλες χώρες και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι τελευταίες πρόοδοι που σημειώθηκαν εδώ και ποια είναι τα μέτρα που προτείνεται για την μη διάκριση κατά τον Ρωμά ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι η αντίδραση ορισμένων ε, Σέρβων πολιτών για τη σύλληψη του Μπλάντιτ ε, συνιστά απόδειξη για το σένος, το κουράγιο που επέδειξε η κυβέρνηση. Άρα θα πρέπει να δούμε και την άλλη οπτική γωνία, την άλλη όψη του νομίσματος. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε όλο το χρόνο του κόσμου μέχρι το 12.30. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη χρονολογική σειρά. Καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που μας ευχαριστείτε και όσον αφορά το θέμα του Μπλάντιτ, θα ήθελα να πω τα εξής. Ε, μην ξεχνάτε ότι η διάλυση της Ιγκοσλαβίας με όλα τα προβλήματα, γιατί πρόκειται για έξι χώρες και 50.000 Σέρβους που εκαθαρίστηκαν από την ε, Βοσνία Ερζεγοβίνη, συν τις 2.000 Σέρβους ε, Ρωμά, μη Αλβανούς, οι οποίοι εκτοπίστηκαν από το Κωσυφοπαίδιο. Ε, αν συγκρίνουμε τα 75 εκατομμύρια ανθρώπων έξω από το εκτός από το βλέπετε ότι 15% του πληθυσμού μας τα τελευταία χρόνια εκδιώχθηκαν από τις αιστείες τους χωρίς απολύτως τίποτε. Και τα παιδιά τα οποία βλέπετε στους ε, δρόμους είναι ακριβώς ε, αυτός ο πληθυσμός. Και θα ήθελα επίσης να επισημίσω ότι η Σερβία ε, ασχολήθηκε ε, από μόνη της με το θέμα αυτό των προσφύγων. Ε, με τις δικές της υποδομές δεν υπήρξε κανένα διεθνές σχέδιο, καμία υποστήριξη από τους διεθνείς δωρητές, από διάσκεψη των δωρητών. Ε, εμείς χρειάστηκε να λύσουμε το πρόβλημα μόνοι μας. Τώρα υπάρχουν ορισμένα προγράμματα και θα πρέπει να πω ότι σε σχέση με την κοινή γνώμη δεν είναι περίεργο. Ο πρόεδρος Τάντιτς είπε ότι οποιοδήποτε διαταράσει την ε, ένομη τάξη θα διωχθεί. Και αυτό δεν είναι μόνο κομμάτι του διεθνού δικαίου, αλλά συνιστά και ηθική υποχρέωση. Γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει για τα αθώα θύματα, για τις μελλοντικέ μας σχέσεις με τις οικογένειες πολιτών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, οικογένειες των θυμάτων. Γιατί ε, τους επόμενους αιώνες θα συνεπάρξουμε με τους Κροάτες, τους ε, Αλβανούς και τους ε, Βόσνιους. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να πράξουμε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Η πλειονότητα των Σέρβων αισθάνθηκε ανακούφιση και όπως είπε ο πρόεδρος Τάντιτς, πραγματικά με τον τρόπο αυτό απομακρύνουμε μια κοιλίδα από τη φήμη μας. Και ε, με τον τρόπο αυτό θα, μας, ε, θα με εμπιστευτείτε μελλοντικά περισσότερο ε, και σας λέω ότι θα κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας για να συλλάβουμε τον στρατηγό Χάτζης. Ε, γιατί και τώρα, αν διαβάσουμε την έκθεση που υπευλήθη από το, για το Συμβούλιο Ασφαλείας του, των Ηνωμένων Εθνών, η Σερβία δεν ε, κάνει ό,τι μπορεί για να συλλάβει τους ε, ε, δύο αναπομείνοντες εγκληματίους πολέμους. Πρόκειται για την έκθεση Μπράμερτς. ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα εδώ και αυτό είναι σημαντικό γιατί ε, ο γνώμων τη προόδου δεν επινοήθηκε για μα, υπέρ ημών, αλλά είναι συνιστά το αντικειμενικό. Τώρα, όσον αφορά το κοσυφομπέδιο, είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε για τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι να είμαστε ευέλικτοι και θέλουμε να είμαστε προβλέψιμοι και αξιόπιστοι ως εταίροι. Αλλά αυτό που λέμε το το, η λύση του, του, Φεβρουαρίου 2008 δεν είναι αποδεκτή από εμά. Πώς μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα, γιατί ήταν μονομερής αυτή η απόφαση της... Ε, ε, οι Αλβανοί στο Κωσοφιοπέδιο δεν θέλουν να κυβερνώνται από το Βελιγράδι. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά και οι μη Αλβανοί δεν θέλουν να κυβερνώνται από την Πριστίνα. Δεν είναι δυνατόν να βλέπω μόνο τη μία πτυχή, τη μία όψη της πραγματικότητας. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την ίδια την πραγματικότητα. Αν θέλουμε να την αλλάξουμε, αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπέρ τη βίας και κανείς πλέον δεν μπορεί να επιθυμεί τη βία. Και αν θέλουμε να αναζητήσουμε μια ειρηνική λύση, θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη και βεβαίως εδώ στην ΕΦΕΤ δεν έχω ούτε την εξουσιοδότηση ούτε είναι ενδειγμένος τόπος να το πράξω αλλά βεβαίως το μήνυμά μου είναι ότι είμαστε δεθειμένοι να συνομιλήσουμε για τα πάντα, για το βόρειο κοσυφοπαίδιο. Ε, επίσης όλα τα θέματα ε, ούτως ώστε να μην είναι μην υπαγωμένη η σύγκρουση αλλά να υπάρξει μια βάση ευημερίας σε αυτό το τμήμα των Δυτικών Βαλκανίων αυτό τον αιώνα αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή η οποία είναι ξεκάθαρη. Μη μας ε, ζητήσετε να κινηθούμε ε, αντίθετα προς το σύνταγμά μας. Αλλά θα βρούμε μια λύση και θα βρούμε μια λύση αν μας τίνεται μια χείρα βοηθείας. Γιατί στο Κοσφόδιο και αναφέρομαι σε δύο εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 300 εκατομμύρια ευρώ ε, εξαγωγών. The stake in making sure ε, και αυτός ε, ε, και πραγματικά εμείς πηγαίνουμε στο σωστό δρόμο. Τώρα, όσον αφορά κάποια άλλα θέματα, ε, υποστηρίζουμε πλήρως τη Γιούλεξ Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο συνέβη τις τελευταίες μέρες όταν η Γιούλεξ εξέδωσε ένα ένταλμα σύλληψης για κάποιον στην Τουρκία, η Ιντερπολ είπε ναι, πρόκειται για ένα αντιθέσει ένταλμα και χθες σε μια σερβική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας ο γιατρός αυτός ο οποίος είναι ύποπτος για εμπορία μεταμόσχευση οργάνων είπε ότι, είμαι, ότι είναι ελεύθερος. Ε, η Γιούλεξ ε, και δεν είναι το σφάλμα της Γιούλεξ. Η Γιούλεξ δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Ε, δεν ισχύει έντολη, το ένταλμα εκτός του, του κοσυφοπεδίου για το υπόλοιπο της Σερβίας, για την Αλβανία, για την Τουρκία, για το Μαρόκο ε, ε, όπου θα γίνουν σημαντικές ανακρίσεις. Ε, δεν, αυτό δεν το λέω κατά της Ε, και το θέμα αυτό είναι σημαντικό. Οι άνθρωποι αυτοί φωνεύτηκαν προκειμένου τα όργανα τους να απολυθούν στη διεθνή αγορά. Πρόκειται για ένα μείζον θέμα, όχι ελάσσον. Ε, δεν θα πρέπει να φροντίσουμε και αυτές και τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Και αυτό ακριβώς ε, ζητούμε. Και εδώ ε, βάζω μια ξεκάθαρη γραμμή. Εμεί στη Σερβία και μπορείτε να δείτε τι δηλώσει του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου κλπ. Ποτέ δεν πολιτικοποίησαμε αυτό το θέμα. Καμία στιγμή δεν το πολιτικοποίησαμε. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ποτέ δεν το εντάξαμε στο διάλογο με την Πριστίνα ή σε πολιτικό επίπεδο. Αφορά τη διεθνή δικαιοσύνη. Τώρα, όσον αφορά την Κροατία, χαιρετίζουμε την ε, ένταξη της Κροατίας και αναφέρατε το Δούναβι. Αυτή τη στιγμή η Κροατία μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ο Δούναβης θα ρεύσει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σερβία και θα ξαναμπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Ρωμανία και στη Βουλγαρία. Και νομίζω ότι δείχνει ότι η Κροατία δεν είναι μόνο κομμάτι της Ευρώπης, αλλά φυσικό κομμάτι της Ευρώπης, φυσικό τμήμα της Ευρώπης. Ε, υπάρχουν ορισμένα άλλα θέματα, αλλά η διμερή σχέση μεταξύ Ζάγκρεπ και Βελγραδίου ε, βελτιώνεται. Και μπορώ να σας δώσω σοβαρά παραδείγματα. Ε, σας έφερε την επίσκεψη στο Βούκοβαρ, κοινά, ε, κοινά σχέδια νοικοδόμηση του Βούκοβαρ και επίσης κάποιες σερβικές επενδύσεις που επιτέλους επιτράπηκαν στην Κροατία στις 22 Ιουνίου για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια θα γίνει μια απευθείας ε, εναέρια σύνδεση μεταξύ Βελιγραδίου και Ντουμπρόβνικ και ε, ορισμένοι θαυμάσιοι άνθρωποι ε, μεταξύ Σερβίας και Σέρβοι και Κροάτες ξανά ντρεύονται μεταξύ τους. This is, I, didn't mean... Δεν και όσον αφορά τη Βοσνία ριζεγοβινη πιστεύω ότι η δήλωση του Τάντιτς σε σχέση με τη Σεμπρένιτσα, στη Σεμπρένιτσα δείχνουν ότι η Σερβία υποστηρίζει την εδαφική ακαιρεότητα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε και θα υποστηρίζουμε κάθε λύση για το ούτως ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν οι τρεις λαοί της Βοσνίας και δεν πρόκειται να υπονομεύσουμε την γραφική ακαιρεότητα τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τώρα, κατά πόσο είναι σοβαρέ μεταρρυθμίσει στη Σερβία ή όχι. Ε, ε δεδομένη προέλευσή μου, νομίζω δεν έχει νόημα να σα πω ναι είναι. Είχαμε 17 δισεκατομμύρια ευρώ ξένων επενδύσεων και έχουμε τρεις συμφωνίες, μία από αυτές ένα δις επενδυτών από το Βέλγιο, την Ορβηγία και την Ιταλία στη χώρα μας, κάτι το οποίο δεν θα έκαναν εάν ε, θεωρούσαν το θα είμαστε σοβαροί. Και εγώ είμαι περήφανος γιατί δεχτήκαμε την γαλλική αντιπροσωπεία ε, ε, σε σχέση με τη, με, Μισλέ και είπαν ότι επισκέφθηκαν τις, τα εργοστάσια μας και είπαν ότι είναι τα πιο παραγωγικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα, σαν αφορά τους Ρωμά, και εγώ είμαι πρόεδρος του Συμβουλίου για την ένταξη των ε, Ρωμά. Είναι ένα ηθικό ζήτημα. Εμείς οι Σέρβοι στην Ευρώπη δεν μπορούμε να αποδεχθούμε το γεγονός ότι μια ομάδα ανθρώπων έχουν ε, κατά 15-20 χρόνια χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής από τους υπολείπους. Ε, το 70% των Ρωμά ζουν, διαβιούν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής. Επίσης το ζήτημα των προσφύγων και των ετούντων άσυλο. Συνάντησα την κυρία Γιάροκα από την Ουγγαρία και συζητήσαμε για την πλατφόρμα που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή και τη στρατηγική που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο. Η Ρωμά είναι οι μόνοι Ευρωπαίοι, πράγματι όπως μας λένε ορισμένοι αρχηγοί Ρωμά, που βεβαίως αποτελούν μειονότητα παντού, σε όλες τις χώρες. Άρα η πατρίδα τους είναι η Ευρώπη. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Για πρώτη φορά εξασφαλίσαμε να έχουμε θετικές ε, διακρίσεις ε, για τουλάχιστον 100 φοιτητέ που φοιτούν δωρεάν στα πανεπιστήμια μας. Επίσης προσπαθούμε να κρατήσουμε τους μαθητές γραμμά στα σχολεία Επίσης, είναι πιο αποτελεσματικό να επιλύεται το πρόβλημα εκεί που, που υπάρχει, αντί να παίζουμε ένα είδος πινκ-πονγκ με τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Και στη Σερβία πάντοτε λέμε ότι το μέλλον των ανθρώπων, των Ρωμά, βρίσκεται στη Σερβία. Και θα θέσουμε στη διάθεση στοιχεία σε σχέση με το τι κάνουμε. Στις 22 Ιουνίου με τον κύριο Μιρέλ από την Επιτροπή Διεύρυνση. θα έχουμε μια ημερίδα για την ένταξη των Ρωμά στη Σερβία. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι δεν υπάρχουν καθόλου περιστατικά βίας κατά τον Ρωμά, ελάχιστα περιστατικά. Εγώ είδα ένα παιδί το οποίο το είχαν δύρει και πριν από τρεις εβδομάδες ο δήμαρχος ε, του Βελιγραδίου ε, το καλωσόρισε όχι μόνο αυτό το παιδί θύμα αλλά και το παιδί από το Βελιγράδι που το προστάτεψε λέγοντας ότι αυτό το παιδί που προστάτευσε το μικρό Ρωμά είναι ο αληθινός ήρωας του Βελιγραδίου. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Ε, ελπίζω ότι κάλυψα τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω ότι κάποια από εσά τουλάχιστον θα έρθετε στο Βελιγράδι, γιατί όπως είπε ο, ο Άγιος ε, ε, το να βλέπει κανείς με τα μάτια του <laughs> σημαίνει ότι πιστεύει. Λοιπόν, η επόμενη συνάντηση θα γίνει στις 21 Ιουνίου στις 9 το πρωί εδώ στις Βρυξέλλες.